Καλημέρα σας. Λοιπόν, προσπαθήστε όσο μπορείτε πιο γρήγορα να βρείτε τις θέσεις σα, γιατί η ώρα έχει πάει 9 και μας περιμένει μια πολύ μεγάλη μέρα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Και πριν ε, οτιδήποτε άλλο θα ήθελα να σας πω ότι χτες ε, δεν συζητήθηκαν οι αφισβητούμενες συστάσεις, οπότε χρειάζεται χρόνο απόψε στου συντονιστές αν δεν είμαστε πάρα πολύ φλίαροι, έχουμε ε, υπολογίσει ότι στις 6 παρατέταρτο μπορεί να αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ, όταν παίρνετε το λόγο, θυμηθείτε να σταματάτε κιόλας. Δηλαδή, όσο γίνεται, να μην μακρύγορείτε. Έτσι θα αξιοποιήσουμε τη μέρα. Λοιπόν, ε, αποφάσεις των συντονιστών έχουν ως εξής. Εγκρίθηκε η μερίσια διάταξη του Φεβρουαρίου και τα αιτήματα για αργότερα. Ε, συμπεριλήφθησαν όλες ε, όλα τα αιτήματα ε, των πολιτικών ομάδων εκτός από την αναφορά 0051 για την Ντονιάνα που πήγε το Μάρτιο και μετά από αίτημα των σοσιαλιστών αντικαταστάθηκε από την 841. Η 073 θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του Μαρτίου και θα προσκληθεί και ο Δήμαρχος του Μαραθώνος ε, στη συνεδρίαση αυτή. Για τη 0841 ήταν επίγον να αποφασιστεί και αποφασίστηκε να ζητηθούν πληροφορίες από τις Γαλλικές Αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι υπόλοιπες αμφισβητούμενες συστάσεις θα συζητηθούν σήμερα, όπως σας είπα σας παρακαλώ ε, δείξτε μια αυτοσυγκράτηση όσο γίνεται για να μπορέσουν να συνδυάσουν ε, και οι συντονιστές κατά τις 6 παρατέταρτο όπως σας είπα. Ελπίζω. Για τα θέματα Β ε, θα συμπεριληφθούν στα γραπτά ε, συμπεράσματα για την ε, αποστολή στη Γερμανία ασχολήθηκαν οι συντονιστές με το πρόγραμμα και την αλλαγή της σύνθεσης. Παρακαλώ οι σύμβουλοι μην κάνετε τόση φασαρία. Εδώ αριστερά, λίγο πιο ήσυχα σας παρακαλώ. Everybody is looking at you at this moment. Και όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους επάνω σας. Ε. Προσπαθείτε να καθίσετε γρήγορα. Fine. So, The second fact Τι έλεγα λοιπόν, δεύτερη διερευνητική ε, αποστολή ε, στο πρώτο εξάμεινο του 2018 θα είναι διήμερη το Μάιο στην Αμόχωστο. Δημόσια κρόαση για το Brexit, 1η Φεβρουαρίου το απόγευμα. Και έχει ε, συνδιοργάνωση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΑ. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Δημόσια αγρόαση, ακρόαση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ε, σε συνεργασία με την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Σημείωσαν χθε το σχέδιο ημερήσιας διάταξη των Το ερευνητικό πρόγραμμα τώρα αποφασίσαμε να παραμείνει ο κατάλογος όπως είχε προταθεί στο παρελθόν. Αλλαγή ζητήθηκε από τους πρασίνους για να αντικατασταθεί μια μελέτη από τη μελέτη για τη σήμανση τροφίμων, ζωοτροφών και καλλιντικών. Εγκρίθηκε αυτό το αίτημα. Προφορική ερώτηση τώρα αποφασίστηκε να κατατεθεί μαζί με ψήφισμα για τα θέματα της ακρόασης για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ε, προσωρινή επισφαλή εργασία. Χάρη σε εσάς κυρία Βαγίνα σώζετε την τιμή της Επιτροπής μας γιατί αποφασίσατε να πάτε στο Περού, στη Λίμα για το θέμα των αναφορών και ε, εκεί θα προεδρεύει η κυρία Ρενάτε Βέμπερ στην αντιπροσωπεία που θα είναι σε επαφή και με τη δική μας γραμματεία. Τουλάχιστον δύο έχουμε που μπορούν να μας ενημερώσουν για την διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ και πάλι. Πρόγραμμα εργασίας και εκθέσεις για το 2019 Κλήθησαν οι συντονιστές να υποβάλουν προτάσεις μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, πάντα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Και επίσης ε, γκρίθηκε η πρόταση να έρθουν κάποια μέλη να παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες τους στην Επιτροπή όταν είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Φάτκα. Ε, ε, αυτό το, θέμα το φορολογικό έχει ε, αναβληθεί γιατί δεν έχει απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χτες αποφάσισαν οι συντονιστές να παραμείνουν σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσουμε ταχεία απόκριση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να επανέλθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας απαντήσει για το τι μέλη και πώς πρέπει να συνεχίσουμε. Τελικά οι συντονιστές επίσης σημείωσαν και κάποια ενημερωτικά στοιχεία ο πλήρης κατάλογος θα δοθεί γραπτός. Αυτά από συντονιστές. Ας προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία, αλλά προηγουμένως να σας κάνω και μερικές ανακοινώσεις. Σήμερα, γύρω στις 10.30, θα έχουμε αντιπροσωπεία επταμελή από τη Βολή του Μαρόκου που θα έρθουν γιατί ενδιαφέρονται να δουν τη λειτουργία της Επιτροπής Αναφορών ε, Πώ λειτουργεί και εργάζεται μια επιτροπή σαν τη δική μας και θα ακολουθήσει και γεύμα που θα παρατεθεί, όπου μπορείτε να έχετε συζητήσει και επαφέ κατά τη διάρκεια του γεύματος μαζί του αν ενδιαφέρεστε. Επίσης, έχουμε και ε, πράσινους ε, αγρότες από την Αυστρία ε, που ενδιαφέρονται πολύ να δουν πώς λειτουργεί η Επιτροπή μα. Λοιπόν, Έχετε τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε. Σας αφήνω λίγο χρόνο να τις βρείτε. Don't <laughs> <laughs> get that. Don't get that. You started. Λοιπόν, καλωσορίσατε κύριε Βίλαντ. Ωραία, βάλατε και την κάρτα σας στο μηχάνημα, τέλεια. Προχωρούμε λοιπόν και ψηφίζουμε. Σχέδιο συνοπτικού ψηφίσματος ε, για την προστασία των μειονοτήτων και την απαγόρευση των διακρίσεων στα, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αιτιολογική αναφορά 3. Ψηφί υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 6 το πρώτο τμήμα. Ε, Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Citation 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τελογική αναφορά 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη τώρα, σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Α, όχι, όχι, καταπίπτει. Καταπίπτει, έχετε δίκιο. Ωραία. Αιτιολογική αναφορά, ό Επίση σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο καταπίπτει. Για να δούμε τώρα που θα πάμε. Στην παράγραφο 11 ψηφί περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Το πρώτο τμήμα. Α, είναι χωριστή ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται έλεγχο. Παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Και τελειώνει τώρα. Τι έγινε. Ε, κύριε Παγίνα, κάτι έγινε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, ξανά αρχίζει τώρα. Σεσίλια, δεν λειτουργεί το μηχάνημα της κυρίας Βαγίνα. Try another. Καλά, δοκιμάστε το διπλανό. Εγκρίθηκε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα στην κατατμήματα ψηφοφορία, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές. Και αυτό θέλει έλεγχο. And let's Πέρας. Εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το υπόλοιπο καταπίπτει. Και θα πάμε τώρα στην παράφο 14. Καταπίπτει είπαμε αφού απερίφθη το προηγούμενο. Λοιπόν, παράγραφος 14, σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 15, πάλι σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 16 Ε, χωρίς την ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα οι κατατμήματα, το split, ε, δύο τμήματα έχουμε υπέρ του πρώτου κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρα καταπληκτούν τα υπόλοιπα. Παράγραφος 17 λοιπόν υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονική επαλήθευση για την παράγραφο 17 πέρας εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά παρακαλώ καλά που το ελέγξαμε έχουμε και προφορική τροπολογία εδώ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Παράγραφος 18 υπέρ κατά αποχές και αυτό θέλει έλεγχο παρακαλώ. Αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 19 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τελική ψήφος ηλεκτρονικά τώρα, τελική ψηφοφορία για το σύνολο. Πες. Εγκρίθηκε. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Thank you for that. And we move to the opinion on the Μπορούμε τώρα λοιπόν να περάσουμε σε γνωμοδότηση ε, μια κοινογιάρα και εδώ για την πρωτοβουλία πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ. Πριν ξεκινήσουμε και δώσουμε το λόγο στο Γιάρεκ, θα ήθελα να ζητήσω από όσους έχουν σκοπό να εγκαταλείψουν την αίθουσα να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα ε, γίνεται το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε αυτή την αναθεώρηση της, πρωτοβουλίας, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ε, Πολιτών και να σας πω πως τη βασική έκθεση θα την προετοιμάσει η ΑΦΚΟ ε, και μετά θα συνεχίσει με το θέμα αυτό με τη δεύτερη έκθεση ε, η ΚΑΛΤ. Το Σεπτέμβριο του 2017 εγκρίθηκε μια, ένα ψηφίσμα με μια πρόταση που έχει σκοπό να αναθεωρήσει εκ αυτόν τον ε, κανονισμό έτσι ώστε να καλύψουμε το βασικό μας στόχο που είναι αυτή η πρωτοβουλία να είναι πιο εύκολη, λιγότερο δυσχερής, πιο φιλική προς τον οργανωτή έτσι ώστε να μπορούν ε, οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν όλο το γάμα δυνατοτήτων αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών γιατί είχε αρχικά σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο που θα ε, τροφοδοτήσει τη συζήτηση που θα φέρει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στους θεσμούς αυτής που θα τους δώσει την αίσθηση της συμμετοχής και χαίρομαι γιατί βλέπω πως η Κομισιόν με την πρότασή της ε, παρουσιάζει κάποια στοιχεία τα οποία ε, είναι παρόμοια με αυτά τα οποία παρουσιάσαμε εμείς πέρσι τον Ιούλιο. Οπότε αυτό το βρίσκω πολύ ικανοποιητικό και αν το εξετάσουμε με λεπτομέρειες θα δείτε πως η αποκλειστική αρμοδιότητα ε, της δικής μας Επιτροπής καλύπτεται από τον κανόνα 54 και εξακολουθεί να ισχύει. Τώρα η πρόταση της Κομισιόν τι λέει. Δεν θα μπω σε όλα τα σημεία της πρότασης αυτής, θα σταθώ στα βασικά. Καταρχήν, βελτιώσεις στην καταχώρηση με τη δυνατότητα της μερικής καταχώρησης ε, πρωτοβουλειών. Επίσης θα εισαχθεί ε, μια, ε, η ιδέα μιας πλατφόρμας online από την ε, Κομισιόν την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όσοι οργανώνουν μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Επίσης, μια, ένα σύστημα συλλογής υπογραφών κεντρικό, ηλεκτρονικό, το οποίο θα το τρέχει η Κομισιόν και η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής θα πέσει στα 16 έτη. Ελπίζουμε πως με τον τρόπο αυτό θα έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία για τον κύκλο ζωής ε, μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και όσοι προωθούν μια τέτοια εκστρατεία θα μπορούν να επιλέγουν από ποια ημερομηνία και μετά ξεκινά να τρέχει η προθεσμία συλλογής υπογραφών. Ελπίζουμε πως το καινούργιο αυτό ε, σύστημα θα βοηθήσει με, την, ε, με το θέμα των υπογραφών και τις υποχρεώσεις εκεί και ελπίζουμε πως θα γίνει πιο διάφανο και πως επίσης θα ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη μέσω αυτής της δυνατότητας. Οπότε ε, ελπίζουμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη διαφάνεια και σε επίπεδο χρηματοδότησης αυτών των ε, πρωτοβουλειών. Όλα αυτά τα σημεία όντως προσπαθούν να πετύχουν το στόχο μας που είναι να ξεδιπλώσει την πλήρη γκάμα δυνατοτήτων που έχει αυτό το εργαλείο, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και νομίζω ότι στην πρώτη δική μας γνωμοδότηση πέρσι ε, είχαμε παρόμοια ε, σχόλια και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έλαβε υπόψη. Στο άρθρο 14 για τις δημόσιες ακροάσεις με χαρά μπορώ να σας πω πώς γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι ε, ε, αποκλειστική αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε Και θέλω να πω και δύο λόγια για το πώς αντιμετωπίζω εγώ προσωπικά την ε, πρόταση. Όπως σας είπα προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της αυτή έχει ε, συμπεριλάβει πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία όμως πιστεύω πως μπορούμε να εμπλουτίσουμε με τις δικές μας. Λοιπόν, καταρχήν, η αποκλειστική αρμοδιότητα για τις ακροάσεις. Είναι δικό μας θέμα, ναι, αλλά ε, στο σχέδιο γνωμοδότησης νομίζω ότι θα πρέπει να το διευρύνουμε και σε επίπεδο διαδικαστικό και σε επίπεδο τεχνικό τη στιγμή τη κατάθεση και επιστοποίηση μια τέτοια πρωτοβουλία. Η πρόταση πάντω έχει μερικά πολύ θετικά στοιχεία. Είναι καλή ιδέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής με τη διατύπωση ε, που λέει μια εξισορροπημένη ακρόαση, δηλαδή όπου θα εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερούμενοι και πιστεύω ότι εμεί θα πρέπει να του οργανώνουμε και να προσκαλούμε τι ακρόασει αυτέ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι εκπρόσωποι των τριών θεσμών, δηλαδή του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και άλλων θεσμών και γνωμοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, και εδώ θέλω να προσθέσουμε και τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους, ε, πιστεύω θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία κάθε στιγμή να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ακροάσεις. Θα πρέπει να τους προσκαλούμε και πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε επίσης και την ορατότητα που έχουν κάποιες τέτοιου είδους πετυχημένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ε, πολιτών. Θα πρέπει να φαίνονται, να τις βλέπει το κοινό. Και η πρότασή μου είναι να γίνεται και μια συζήτηση στην Ολομέλεια ενδεχομένω. Όταν κάποια τέτοια πρωτοβουλία ε, κρυθεί πετυχημένη και ενδεχομένως να συνοδεύεται η συζήτηση αυτή και από ψήφισμα στην Ολομέλεια. Επίσης, είναι σημαντικό τα οδηπορικά ε, προς την ακρόαση να καταβάλλονται στους οργανωτές της πρωτοβουλίας και εφόσον γίνεται στις ε, ακροάσεις που κάνουμε εμείς, γιατί να μην γίνεται και για τις ακροάσεις που οργανώνουμε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Να τους καλύπτουμε λοιπόν τα οδηπορικά. Επίσης, φυσικά σημεία επαφή στα κράτη-μέλη να υπάρχουν για να προσφέρουν κατευθυντήριες γραμμές ε, στους οργανωτές. Μην ξεχνάμε πως δεν χρησιμοποιούν όλοι ακόμα το ίντερνετ. Να εξασφαλίσουμε λοιπόν πως το ευρύτερο κοινό γνωρίζει πως υπάρχει το εργαλείο και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να υπάρχει και αυτή η φυσική παρουσία κάπου. Τέλος. Θα ήθελα να θέσω και ένα θέμα που είναι πραγματικά καυτό και το οποίο το είχα συμπεριλάβει και στην πρώτη μου νομοδότηση πέρσι. Προφανώς υπάρχει κάπου σύγκρουση συμφερόντων και νομίζω αυτό θα το δούμε αν εξετάσουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Αρμοδιότητα Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάσει το παραδεκτό μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και για να την καταχωρήσει και μετά να δώσει και νομοθετική συνέχεια. Άρα λοιπόν είναι όλα στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θέλει να συνδιοργανώνει και τι ακροάσει. Μα κατά τη γνώμη μου, εδώ υπάρχει ε, προφανή σύγκρουση συμφερόντων και η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει να δοθεί αλλού. Δεν ξέρω πώ αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί δεν βλέπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εύκολα να παραδίδει τα όπλα στο σημείο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εμεί θα πρέπει να τονίσουμε πω κάτι πρέπει να κάνουμε σχετικά για να ξεπεράσουμε το θέμα αυτό, να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να μην συγκεντρώνονται οι αρμοδιότητες όλες στα ίδια χέρια. Πολύ λογικό. Για να δούμε τι θέλουν να πούνε οι συνάδελφοι. Έχουμε κάποιους σκιώδες εδώ. Κυρία Μίτση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που είναι βραχνή η φωνή μου. Σίγουρα αυτή η πρωτοβουλία έχει ήδη καθυστερήσει έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Δεν νομίζω ότι υπήρξε επαρκώς επιτυχή. Δεν πιστεύω ότι έλαβαν οι πολίτε όλα τα δικαιώματα και όλες τις πληροφορίε που έπρεπε να λάβουν. Έχουν προταθεί διάφορες αλλαγέ, πιστεύω θετικέ. Πιστεύω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, η πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά ώστε να μετατραπεί σε μια επιτυχή άσκηση, σε ένα επιτυχές εγχείρημα και όχι σε σπατάλη χρόνου. Να μην επανέλθουμε σε μερικά χρόνια με τα ίδια προβλήματα. Τα δικαιώματα των πολιτών πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν περαιτέρω, πιστεύω. Να δούμε αποτελέσματα και επίσης ε, πρέπει να υπάρξει κάποια εγγύηση κατά των ε, επαχθών κανόνων νησιά, οι οποίοι θα πρέπει να μετατραπούν σε πιο φιλικά μέτρα. Αλλιώ η κατάσταση δεν θα αλλάξει. Για να είμαι σύντομη, θα επικεντρωθώ σε αυτά που εξέτασα εγώ όσον αφορά την εκθέση αυτή. Κάτι σημαντικό, απαιτούμενος αριθμός υπογραφών. Αυτή τη στιγμή είναι ένα εκατομμύριο υπογραφές, αλλά τι γίνεται αν έχουμε 800.000 υπογραφές, τις αγνοούμε. για να είναι αποτελεσματική η πρωτοβουλία ως προς το κόστος αλλά και δημοκρατική θα πρέπει να βρούμε μια λύση για την περίπτωση που έχουμε μεγάλο αριθμό υπογραφών χωρίς να έχει ε, υπερβεί το 1 εκατομμύριο. Η συλλογή των υπογραφών, η Επιτροπή λέει ότι πρέπει να καταμετρώνται οι υπογραφές στο κράτος μέλος της υπηκότητας, αλλά τι γίνεται με όσους ζουν στο εξωτερικό. Είναι, είναι διαμένοντας ένα άλλο κράτος μέλος, τους αγνοούμε. Επίσης καλωσορίζω το νέο άρθρο για την ενημέρωση και την αρρωγή όπως προβλέπεται από την Κομισιόν για την οργάνωση της CCI και ειδικότερα τις νέες διατάξεις για το online μετρό και τις υπηρεσίες μετάφρασης που θα παράσχει η Κομισιόν. Αλλά θα πρέπει να πούμε πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει ακριβώς ε, ενημέρωση, αρρωγή και μετάφραση η προαπέτηση ε, εγγραφής ε, για τη CCI δημιουργεί τρία ζητήματα. Το εύρος του αντικειμένου των πρωτοβουλειών, η εγγραφή και η εξήγηση των απορρίψεων ε, εγγραφής. Αυτά δεν εξετάζονται επαρκώς, είναι πραγματικά προβλήματα τα οποία συναντούν οι πολίτες. Το επόμενο στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθούμε είναι η ομάδα των ε, διοργανωτών. Ε, πρέπει να εξετάσουμε κάποιες καταστάσεις, ειδικότερα όταν νομικά πρόσωπα θέλουν να συμμετέχουν στην ομάδα των διοργανωτών. Και τι γίνεται με τις ευθύνες και τις κυρώσεις και πώς όλα αυτά επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες των πολιτών. Και εδώ χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις. Καλωσορίζω λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν να, παρασχεθεί στους διοργανωτές η ευελιξία να αποφασίζουν αυτοί πότε θα αρχίζουν τη συλλογή των υπογραφών. Αυτό είναι μια καλή παρατηρήση. Αλλά το γεγονό τώρα ότι οι διοργανωτές θα μπορούν να τροποποιήσουν την πρωτοβουλία ή να την ε, καταχωρούν ε, εν μέρη στην Κομισιόν είναι πράγματα που χρήζουν περισσότερων εξηγήσεων. Αυτές είναι κάποιες αρχικές μου σκέψεις. Είμαι βέβαιη ότι μόλι κυκλοφορήσει η γνωμοδότησή της ΠΕΤΗ θα έχω να κάνω και άλλα σχόλια. επίση. καλώ ορίζω το τελευταίο που είπατε. Πιστεύω ήταν ε, πολύ εύστοχο. δίδονται υπερβολικά πολλέ εξουσίε στην Κομισιόν πιστεύω Χρειαζόμαστε μία προσέγγιση περισσότερων ενδιαφερομένων. Ε, θα συνεργαστούμε με τον ε, εισηγητή για όλα αυτά. Ε, πρόεδρο χαίρομαι όταν ακούω για τόσο επικοδομητική συνεργασία που ξεκινάει αμέσω. Κύριε Μαριά, σκέφτεστε το ίδιο. Κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ τον συνάδελφο Βαλέσα, να συγχαρώ τον συνάδελφο Βαλέσα για την έκθεσή του. Θα ξεκινήσω με μία παρατήρηση ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ουσιαστικά είναι ένα σύστημα συμμετοχικής δημοκρατίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι την αντιπροσωπευτική δημοκρατία μέσω της εκλογής των Ευρωβουλευτών οι οποίοι και ενεργούν για λογαριασμό των ευρωπαϊκών λαών και για λογαριασμό των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν η διαδικασία πρέπει να απευθύνεται στους πολίτες, πρέπει να μην έχει γραφειοκρατικά στοιχεία και πρέπει να μπορούν οι πολίτες να εκφραστούν άμεσα. Διότι αν μπαίνουν εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία συμμετοχικής δημοκρατίας αντιλαμβάνεστε ότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός της ίδιας της συνθήκης. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα σύγκρουση συμφερόντων στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται η Επιτροπή μέσα σε όλο το σύστημα αυτό. Και είχα την ευκαιρία να μιλήσω στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απευθυνθώ και προς τον κύριο Τίμερμανς και να του πω ότι θα πρέπει να μην έχει τόσες αρμοδιότητες η Κομισιόν. Διότι υποτίθεται ότι οι πολίτες συμμετέχουν άμεσα, μαζεύουν υπογραφές με στόχο να πείσουν την Κομισιόν να αναλάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Άρα δεν μπορεί όλη την προετοιμασία, τον έλεγχο αν η αίτηση είναι σωστή, αν οι συμμετέχοντες είναι πάνω από ένα εκατομμύριο, αν προέρχονται από συγκεκριμένα κράτη-μέλη, όλη αυτή την γραφειοκρατική διαδικασία και τον έλεγχο δεν μπορεί να τον αναλάβει η Κομισιόν η οποία θα δει αν η πρωτοβουλία είναι νομικά και θεσμικά σωστή και εν συνεχεία θα την αποδεχθεί προκειμένου μετά η ίδια να αναγκαστεί να προχωρήσει σε σύνταξη ε, μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Είχα προτείνει λοιπόν ότι όλη αυτή τη διεργασία από θεσμικής πλευράς πρέπει να την αναλάβει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Ένα τελείως διαφορετικό όργανο στο οποίο θα απευθύνονται όλες οι αιτήσει, θα κρίνονται αν είναι νόμιμες ή όχι και αν είναι νόμιμες θα αναλαμβάνει το ρόλο της μετά η Κομισιόν η οποία τι πρέπει να κάνει, πρέπει να συντάξει την νομοθετική πρωτοβουλία. Επομένως, πολύ περισσότερο ισχύει η παρατήρηση του κυρίου Βαλέσα ότι δεν μπορεί να μπει και στο κομμάτι των δημοσίων ακροάσεων κομισιών. Θα έλεγα λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα και πολιτικό ότι καλό θα είναι να ε, διαχωρίσει τη θέση της Κομισιόν από αυτή τη διαδικασία, διότι είναι το όργανο στο οποίο απευθύνονται οι πολίτες και ζητούν κάτι. Αλλά δεν μπορεί να ελέγχει η Κομισιόν όλη τη διαδικασία αυτή των πολιτών. Τώρα, στα άλλα σημεία ε, οπωσδήποτε διευκολύνεται η διεργασία διότι είδαμε ότι είχαμε μια ολόκληρη κινητοποίηση των πολιτών για την TTIP. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση των πολιτών μέσω της πρωτοβουλίας για το θέμα των, του νερού ε, που, δεν, που είναι ένα δημόσιο αγαθό, δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Και είδαμε ότι όλα δεν πήγαν τόσο καλά. Επομένως το ότι αλλάζει ο κανονισμός και γίνονται σημαντικές αλλαγές εγώ το θεωρώ στη θετική κατεύθυνση. Και πρέπει να δούμε μετά τι λεπτομέρειε. Δηλαδή, πρώτον, ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Οι πολίτε στα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά του. Κάποιο πρέπει να του ενημερώνει. Αυτά τα φυσικά σημεία επαφή, όπω λέγονται, η ενημέρωση είναι κάτι το σωστό. Το ότι πρέπει να δοθεί μια τεχνική βοήθεια στου διοργανωτέ, το θέμα τη ε, μετάφραση, το θέμα ε, ορισμένων διευκολύνσεων, οπωσδήποτε είναι σημαντικό ε, και νομίζω ότι είναι προ την σωστή κατεύθυνση. Σε σχέση με αυτό που είπε η συνάδελφο η κυρία Μίτση, να ότι η πρωτοβουλία πολιτών είναι για τους πολίτες. Επομένως οι legal entities, δηλαδή νομικοί, όργανα νομικά ή νομικά πρόσωπα, θα βοηθήσουν. Δηλαδή μια κίνηση πολιτών, παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει αλλά δεν μπορεί να υπογράφει διότι είναι σαφής η συνθήκη. Πρόκειται για συμμετοχική δημοκρατία πολιτών και όχι η συμμετοχική δημοκρατία legal entities, δηλαδή NGOs κλπ. Τα NGOs μπορεί να βοηθήσουν, αλλά την υπογραφή θα την κάνουν τα μέλη τους ατομικά. Το αν θα έχουν ε, μια στήριξη στην όλη διαδικασία είναι ένα άλλο θέμα. Επομένως, για να μην μακρηγορούμε, το θέμα της διαφάνειας το θεωρώ σημαντικό και πιστεύω ότι πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Για μένα αυτό είναι κυρίαρχο, για να μπορούν οι πολίτες να διευκολύνονται. Η ελάχιστη ηλικία 16 έτη το θεωρώ μια σημαντική κατάκτηση, ένα άνοιγμα παιδευτικής διαδικασίας προς τους ίδιους τους πολίτες και τους νεαρούς οι οποίοι στην πορεία θα είναι οι μελλοντικοί πολίτες στα κράτη-μέλη τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό και θα έχουμε πολύ ωραία συνεργασία εδώ. Ε, ευχαριστώ για την συνεισφορά σας και τώρα ο λόγος είναι για τον κύριο Τερή Καμπράς. Thank you. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίσης και εσάς κύριε Βαλένσα και τους υπολείπους συναδέλφους και ηγητές, με τους οποίους συμφωνώ απολύτως με όλα όσα υπόθηκαν. Μια που είμαι και εγώ σκιώδη σύγητης αλλά και για το ίδιο θέμα στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, όλο σκιώδη με βάζουν. Καμιά έκθεση δεν παίρνω. Το πρόβλημά μου είναι ότι μήπως ζω και καμιά σκιώδη ζωή. Λέω τώρα. Να το σκεφτώ. Γιατί δεν έχω χρόνο για πραγματική ζωή. Δεν μπορώ να, να, να ζω στη σκιά συνέχεια. Λοιπόν, επειδή είμαι σκιώδη και στην Αύκο, θα μου επιτρέψετε να επεκταθώ ε, σε αυτό το θέμα από τη σκοπιά των επιχειρημάτων της πολιτικής μου ομάδας. Έχουμε βελτιώσει, σημείωσα 13, μην ανησυχείτε, δεν θα το το σου όλες. Ε, είναι βελτιώσεις μέχρι εκεί θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε ε, μερικά θέματα πολύ σημαντικά. Τέσσερα είναι αυτά. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κρατάει πολύ στενό. Και ε, θα πρέπει ε, να ε, γίνει μια πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλία σε σχέση με τις συνθήκες. Εμείς προτείνουμε να συμπεριληφθούν όλοι οι ε, στόχοι, όλη η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και να είναι ε, της τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να κάνει προτάσεις για μια νέα νομοθεσία για την κατάργηση κείμενης νομοθεσίας ή τροποποίηση κείμενης νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για ε, τροποποίηση των συνθήκων. Δηλαδή θέλουμε λίγο να διευρυνθεί η τροποποιηση κειμενη νομοθεσιας στην ευρωπαικη που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, συμφωνώ πολύ με του συναδέλφου ότι χρειαζόμαστε κάποιο ανεξάρτητο φορέα να κάνει ε, το νομικό έλεγχο για την καταχώρηση. Δεν ξέρω αν είναι ο συνήγορο του πολίτη, ο διαμεσολαβητής ή οποιοδήποτε άλλο. Με χαρά να το συζητήσω αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά χρειάζεται κάποιο ανεξάρτητο όργανο. Το είπε και ο κύριο Βαλένσα πάρα πολύ σωστά και επέμεινε σε αυτό. Σα ευχαριστώ. Τρίτον, η παρακολούθηση. Ε, αυτό είναι η ουσία του θέματο. Γιατί ε, αν κάνουμε καταπληκτικά πράγματα χωρί να τα ολοκληρώνουμε, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Η ε, συνέχεια λοιπόν που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουν γίνει προτάσεις και αλλαγές. Εμείς προτείνουμε να διευκρινίσουμε ότι εξορισμού περιμένουμε ε, πρόταση για νομοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ενίσχυση της διατύπωσης έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγεί τους λόγους ε, στην περίπτωση που αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε δράση. Και το τέταρτο είναι η συνέχεια που δίνει και η παρακολούθηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ούτε εδώ έχουμε αλλαγέ. Η ομάδα μα προτείνει συζήτηση στην Ολομέλεια με ψηφοφορία. Έτσι, με ψήφισμα. Με ε, συστάσεις, συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εάν και κατά πόσο χρειάζεται να προταθεί νομοθεσία και συν τη δυνατότητα να υπάρχει ε, πρόταση για έκθεση ιδέας πρωτοβουλία σε περίπτωση που αδρανήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει πιο ενεργή δράση, προτείνοντας συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η θέση των Πρασίνων και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Μια που θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η δυναμική των πολιτικών ομάδων και ισχυρή η θέση μας, της Επιτροπής μας, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσωπικά πιστεύω, αν μου επιτρέπετε, να πω το εξή. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε πραγματικά τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ε, δούνε και Λαβίν. Το θέμα δεν είναι ότι όποιο κερδίζει τα παίρνει όλα. Το θυμάστε το τραγούδι των Άμπα, The Winner Takes It All. Ε, μοιραζόμαστε ευθύνε και καθήκοντα και τελικά την επιτυχία και τη χαρά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ρόντιγκερ. Α, ξεχάσαμε την ευθύντη, η κυρία Εύη. Συγγνώμη, δεν σα είχα δει. Παρακαλώ. Ελεονόρα. Ευχαριστώ, Σεσίλια. Όσον αφορά το θέμα αυτό, ήθελα να παρεμβώ για να επαναλάβω βέβαια και όσα είπαν οι συνάδελφοι και να εκφράσω τη συμφωνία μου. Ήθελα να εστιάσουμε ωστόσο και σε κάποια σημεία που θεωρώ σημαντικά. Η πρώτη, το πρώτο που θέλω να πω αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι με το μονοπόλιο της ε, ως ε, κατέξουσα την νομοθετική πρωτοβουλία διακινδυνεύει ουσιαστικά την ε, ύπαρξη αυτού του εργαλείου. Κατά την απόψή μου λοιπόν είναι απαραίτητο να αλλάξει αυτό, να αλλάξουμε τις συνθήκες ώστε το μέσο αυτό να ενισχυθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Και να μην έχει τη διακριτική ευχαίρεια από νομική άποψη κομισιών όπως έχει σήμερα. Ε, ξεκινώντας τώρα από αυτό, για να μπούμε στην ουσία ε, της πρότασης κανονισμού, ήθελα να υπενθυμίσω ότι κατά την άποψή μας είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η αρχική καταχώρηση μία τέτοια πρωτοβουλίας και το παραδεκτό της πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο πιο ολοκληρωμένο. Θέλω να υπενθυμίσω την απόφαση του δικαστηρίου για το Stop TTIP που είχε προταθεί ε, για τις προπαρασκευαστικές πράξεις ε, μιας νομοθετικής πρότασης και να υπενθυμίσω πόσο απαραίτητο είναι να υπάρχει και τέτοια τήρηση των δημοκρατικών αρχών και των αρχών συμμετοχής όπως ε, ε, εκφράζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό πιστεύω είναι σημαντικό να το υπενθυμίζουμε. Εμείς θα κάνουμε και σχετικές προτάσεις για τροπολογίες. Θεωρώ ότι μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο τροποποίηση του πρωτεύοντο δικαίου τη Ένωση, τη συνθήκη. Αυτό θα πρέπει να. ή μάλλον συγγνώμη, μια τέτοια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία θα πρέπει να αφορά και τροποποίηση των συνθήκων. Η Κομισιόν δεν μπορεί απλά να παρέχει μια αιτιολόγηση όπω συμβαίνει σήμερα. Η αιτιολόγηση απόρρεψη θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τρόπο πιο σαφή. Και τροποποιηση των συνθηκων η κομισιον δεν μπορει απλα να παρεχει μια αιτιολογηση οπω συμβαινει σημερα η αιτιολογηση απορριψη θα πρεπει να τεκμηριωνεται με τροπο πιο σαφη και επισης και η συλλογή υπογραφών θα πρέπει να επεκταθεί για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες ε, στο μέτωπο αυτό. Ε, να επεκταθεί λοιπόν στους 18 μήνες ε, ως χρονικό πλαίσιο. Κατά τα άλλα συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι επί πολλών σημείων. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεργαστούμε εξαιρετικά για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Βαλίνα, θέλετε το λόγο. Όχι. Πολύ ωραία. Το λόγο έχει τώρα ο εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν, ο κ. Μπόγκαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ για όλα τα σχόλιά σα για όλα τις παρεμβάσεις και παρατηρήσεις και ειδικότερα τον εισηγητή και του ε, ισκιώδεις που είχα την ευχαριστήση να ακούσω χθε. Ε, τι συμπεραίνουμε από όλα αυτά. Έχουμε ένα κοινό στόχο που καθιστά το εργαλείο αυτό πιο προσπελάσιμο, πιο εύχριστο αυτός είναι ο στόχος μας τόσο για τους διοργανωτές όσο και για τους ε, υποστηρικτές του. Θέλουμε επίσης ε, το εργαλείο αυτό να επιτύχει όλους τους στόχους ε, και να αποφέρει όλα τα δυνατά αποτελέσματα. Είμαι ευγνώμων προς όσους παρέθησαν έως και 13 βελτιώσεις. Μπορούμε να το δούμε διμερώς και φυσικά και σε αυτό θα εστιαστούμε μαζί Συμφωνώ με τα όσα είπε η Πρόεδρος ότι η συζήτηση αυτή που γίνεται μεταξύ του συνομοθέτη των κρατών μελών στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και θα έχει και τη δική μας συμμετοχή και ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι να υπογραμμίσω πώς βλέπουμε εμείς ε, βάσει του ρόλου μας ε, ως ε, θεματοφύλακα των συνθήκων και βάσει των εξουσιών που μας προσφέρουν οι συνθήκες, ε, τι ρόλο θα έχουμε εμείς. Αυτό ήθελα να τονίσω και να τονίσω επίσης ότι για πολλά στοιχεία ευχαρίστω θα θέλαμε και εμεί να προβούμε σε μεγαλύτερη ανάλυση. Ε, πρόκειται να γίνει μια συνάντηση νομίζω την επόμενη Τρίτη ε, το απόγευμα. Ξέρω ότι, θα γίνει ότι τη διαχειρίζεται η ΑΦΚΟ. Είμαστε στα χέρια λοιπόν εκεί του Κοινοβουλίου. Εκεί θα εξετάσουμε άρθρο προς άρθρο το κείμενο και όσοι ασχολούνται λοιπόν επιστέμενα με αυτό το αρχείο θα καλό να συμμετέχουν και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ε, δυνατό. Το τελευταίο που ήθελα να τονίσω πριν ε, μπω περισσότερο στην ουσία, είμαστε ευγνώμονε που τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο έχουν θεωρήσει ότι ε, το θέμα αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο τη κοινή διακήρυξη με κάποια φιλοδεξία να υιοθετηθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Οπότε αυτό μας δίνει χρόνο να προετοιμάσουμε όλες αυτές τις βελτίωσεις οι οποίες ελπίζουμε να τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2019. 20. Ε, επιτρέψτε μου να αφιερώσω δύο λεπτά για να σας παρουσιάσω τη θέση της Κομισιόν. Έχουμε το θέμα της καταχώρησης και του follow-up. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι ως αξιωματούχος της Κομισιόν και ως πολίτης θεωρώ ότι το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων ε, δεν είναι σωστό να το αναφέρουμε. Μιλάμε και εξουσίε που χορηγούνται στην, χωρούνται στην Κομισιόν από τι συνθήκε. Δεν μπορεί να αναμένει κανεί κάτι περισσότερο από την Κομισιόν. Απλά να τηρεί αυτέ τι εξουσίε. Και αυτό χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα είναι θεματοφύλακα ε, των συνθήκων η Κομισιόν ε, και του υποκειμένου και εκτιμένου. Οπότε πρέπει να δούμε τι περιλαμβάνουν οι εξουσίε τη. Ε, το είπε πολύ καλά ο Αντιπρόεδρο στι 12 Δεκεμβρίου. Οπότε εδώ αναφερόμαστε στην καταχώρηση. Σε κάποια στιγμή η Κομισιόν πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο είναι εντό των εξουσιών τη, εντό των αρμοδιοτήτων τη το να δράσει. Δεν γίνεται αυτό αυτόματα λοιπόν. Αποτελεί αυτόματο, αυτόματη συνέπεια του γεγονότος ότι οι εξουσίες αυτές έχουν κορθεί στην Κομισιόν. Θα ήταν κρίμα λοιπόν σε κάποια φάση αν ε, αποτιμά όλο αυτό κάποιο άλλο, ε, να το αποτιμά διαφορετικά από την Κομισιόν και αυτό να επηρεάσει τη συνοχή και το follow-up. Το άλλο που ήθελα να πω για την παρακολούθηση για το follow-up είναι το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα ούτε της Κομισιόν, να συζητήσουμε κατά πόσο πρέπει να γίνει αλλαγή των συνθήκων. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλία μέσω του κανονισμού ECI. Αυτό είναι βασικό πρωτογενέ δίκαιο. Και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα εμπλακεί και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου σε αυτέ τι συζητήσει, όπω και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Και ελπίζω μέσα από αυτέ τι συζητήσει να διευκρινίσουμε την κατάσταση ώστε να συζητήσουμε όλα αυτά τα σημεία. Τώρα, ε, για την καταχώρηση. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Συχνά λέγεται κάνουμε μια αξιολόγηση και μετά μια καταχώρηση. Ουσιαστικά ε, πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Η αξιολόγηση είναι το βασικό πράγμα και απλά ακολουθεί η καταχώρηση. Οπότε η αξιολόγηση είναι νομική αξιολόγηση. Μόνο όπως προβλέπεται στον κανονισμό αφορά την νομιμότητα της ε, ε, πρωτοβουλίας. Πρέπει να έχει δείχνει συνοχή με το follow-up που γίνεται μετά που απορρέει από το δικαίωμα πρωτοβουλία και επίση τι έχουμε προβλέψει να υλοποιήσουμε μια γρήγορη ταχεία διαδικασία. Διότι η καταχώρηση είναι η αφετηρία και μετά στην Κομισιόν λέμε ότι ε, θεωρητικά ελπίζουμε να καταχωρούνται μερικώ ή πλήρω όλε οι πρωτοβουλίε. Αυτή είναι και η πρακτική τη Επιτροπή Γιούνκερ. Υπάρχει μόνο, μόνο μία πρωτοβουλία. Ε, η Stop Brexit έχει απορριφθεί από τις έξι που από τις 16 που είχαν ε, προταθεί. Αλλά ε, θα συμφωνήσω, πιστεύω και όλοι οι νομικοί ότι δεν ενέπτε ε, στις αρμοδιότητες της Κομισιόν η πρωτοβουλία αυτή. Όλες οι υπόλοιπες ναι. Πώ κάνουμε την καταχώρηση. Προσπαθούμε να γίνεται με γρήγορο τρόπο, το πολύ σε δύο μήνες, άμεση καταχώρηση, άμεση μετάφραση της πρωτοβουλία, ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και φυσικά μετά από αυτό ε, βάλαμε, τε, μετατρέψαμε την περίοδο σε τρει μήνες για να δίνουμε χρόνο στους διοργανώτε να οργανώθουν σωστά και για να ε, βελτιωθούν οι πιθανότητες επιτυχίας, γιατί οι δύο μήνες ήταν αναποτελεσματικοί. Επίσης, η Κομισιόν λαμβάνει μια επίσημη νομική απόφαση ε, κατά τις οποίες μπορεί να προσφύγει κανείς στο δικαστήριο και ξέρουμε ότι έχει συμβεί και αυτό. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Όταν σκέφτεται κανείς τις αναλλακτικές, η προσφυγή λοιπόν των ε, διοργανωτών αν υπάρξει απόφαση μη καταχώρησης ε, είναι ένα δικαίωμα που θέλουμε να δεν αυτό το οποίο έχουμε προβλέψει ως μια επιπρόσθετη δυνατότητα είναι αυτή η συμμετοχική πλατφόρμα που προσφέρει και νομική αρρωγή, η οποία είναι ανεξάρτητη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου γίνεται μια προαξιολόγηση μέσω αυτής της πλατφόρμας της πρωτοβουλίας πριν τη στείλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους λένε ποια είναι η νομική βάση, ε, το εύρος, το πεδίο, οι δυνατότητες και πιθανότητες επιτυχίας και αφού χρησιμοποιήσουν αυτή τη νομική αρρωγή μετά μπορεί να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα εκτιμήσει αν η πρωτοβουλία είναι παραδεκτή, είναι μερικώς παραδεκτή κτλ. Έτσι μέσα σε ένα μήνα δίνουμε πληροφορίες στους οργανωτές οι οποίοι μετά την ενημέρωση αυτή μπορούν να ξεκινήσουν ή όχι. Και λέμε μέσα σε ένα μήνα. Και τότε έχουν και τη δυνατότητα να επαναξιολογήσουν ε, αλλά αυτό εξαρτάται απολύτω από του οργανωτέ, να επαναδιατυπώσουν κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα παρέμβει γιατί εμεί δεν έχουμε σκοπό να ε, του υποχρεώσουμε ε, να επιλέξουν συγκεκριμένο πεδίο ή όχι, αλλά μπορούμε να τους δώσουμε κάποια απάντηση ήδη για το κατά πόσο ε, θα είναι θετική αποκρισή μας σε επίπεδο παραδεκτού κτλ. Τώρα, για τη μερική καταχώρηση είναι μια μεγάλη δυνατότητα που αποτελεί ένα νέο ξεκίνημα. Καταλαβαίνω αυτά που μας λέτε, αλλά επιστρέφοντας στο θέμα, πιστεύω πως εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο εργαλείο αυτό, έχουμε δύο ρόλους, του οποίους μας αναθέτει η συνθήκη. Πρώτα απ' όλα, το να αξιολογήσουμε ή όχι αν πρέπει να δράσουμε και δεύτερον, το δικαίωμα πρωτοβουλίας να νομοθετήσουμε ή όχι, ή να δράσουμε ή όχι και να το εξηγήσουμε βεβαίως ε, και να το τεκμηριώσουμε παρκώς. Και όταν προχωρήσει η συζήτηση στα δύο αυτά στοιχεία θα ήθελα να δώσω κάποια στοιχεία για προβληματισμό για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, μέσα βέβαια στα πλαίσια τα οποία πιστεύουμε πως μας δεσμεύουν. Γιατί υπάρχουν όρια και τα όρια αυτά τα θέτουν οι συνθήκες. Ελπίζω ε, να μακρηγόρησα μένα, αλλά να ήμουν σαφής δε, έτσι ώστε να εξήγησα επαρκώς και να καθησύχασα τις ανησυχίες σας. Ήσασταν απόλυτα σαφής, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Βαλέσα. Για μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που είμαστε τόσο ενωμένοι και χαίρομαι ιδιαίτερα που όλοι ε, ακολουθούμε ε, την ίδια πορεία και Χαίρομαι και βέβαια είμαστε όλοι ενωμένοι, μάλλον κάπως εναντίον της Κομισιόν και η οποία μας απάντησε λίγο πολύ αυτά τα οποία αναμένονταν πως ε, οι αρμοδιότητες περιγράφονται στη συνθήκη και η αποκλειστική αρμοδιότητα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών βρίσκεται και αυτή στη συνθήκη κτλ. Οπότε η δική μας δουλειά θα είναι να τους πείσουμε να παραδεχτούν πως κάτι χρειάζεται να γίνει έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση έτσι ώστε να μην έχει μόνο την απόλυτη εξουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δικαίωμα πρωτοβουλίας των πολιτών για να επιμείνουν στο να ξεκινήσει μια νομοθετική διαδικασία δεν είναι ένα δικαίωμα ότι θα πρέπει να αξιολογείται και να κρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα χρειάζεται ένα αυτόνομο όργανο. Βέβαια είναι διαδικαστικό θέμα και έτσι περιγράφεται στις συνθήκες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά ίσως στο τέλος θα καταφέρουμε να πείσουμε τους εκπροσώπους της Κομισιόν ότι κάτι χρειάζεται να αλλάξουμε εμείς εδώ. Και αυτό θα το θεωρήσω πετυχημένο. Σας ευχαριστώ πολύ και ξέρω πως ε, θα τα πάμε πολύ καλά. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι πεπισμένη ότι αν κάποιο μπορεί να πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό είσαι εσύ Γιάρεκ, Εμπρό λοιπόν. <clears throat> Και σα εύχομαι και στου δύο πολύ καλή και γόνιμη συνεργασία. Κομισιόν και εισηγητή μα σίγουρα κάπου θα καταλήξετε. Να θυμίσω λίγο το χρονοδιάγραμμα μου επιτρέπετε. δημόσια χρόαση θα είναι στις 21 Φεβρουαρίου. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 1η Μαρτίου στις 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ αυτό. Και τώρα να καλωσορίσουμε τους αναφέροντες στην Επιτροπή μας. Έχουμε την ε, αναφορά 89 ε, του 1998. Είναι η αρχαιότερη αναφορά μας αυτή η ιστορική στιγμή που ζούμε. Θα ασχοληθούμε με αναφορές που εκκρεμούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για τα θεσμικά όργανα πέντε συνολικά. Θα δώσω πρώτα το λόγο με χαρά στον David Petrie, ο οποίος είναι ο συντάκτης της αναφοράς της παλαιότερης ακόμα ανοιχτής αναφοράς του Κοινοβούλου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή για την υποστήριξη και την επιμονή της και δεν είναι μόνο η αρχαιότερη περίπτωση, χωρίς καμία αμφιβολία είναι και η μεγαλύτερη περίπτωση μαζικής διάκρισης που βασίζεται σε ε, εθνικότητα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τον Οκτώβριο οι Financial Times δημοσίευσαν μια επιστολή σε σχέση με την απόφαση του αριού πάγου της Ιταλίας του Ιλίου του 2017. Αυτές οι αποφάσεις επανερμηνεύουν προηγούμενες αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκού ε, Ο Άριος Πάγος, ε, το, το δικαστήριο κυρωτικό ε, στην Ιταλία, αρνήθηκε να προβεί σε κάποιες ενέργειες και αμφισβητεί έτσι ότι όλη την ένωμη τάξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξι αποφάσεις έχουμε υπέρ μας. Η πρώτη ήταν το 1998 και η τελευταία το 2008 που αφορά Βελγίδα Νάση Ντελέη που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Ε, η Ιταλία τέσσερις φορές έχει αλλάξει την νομοθεσία τη και πιο πρόσφατα το 2017. Ωστόσο συνεχίζεται η διάκριση. Σας δείχνω σε ένα παράρτημα και σε ένα έγγραφο ε, παραδείγματα με πίνακες και στοιχεία. Α έρθουμε όμως στην υπόθεση της κυρίας Ντελέη. Προσβάλλει και τη συνθήκη και το κύρος ε, του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2008 το ΔΕΚ έθεσε τις αρχές που θα πρέπει ε, να τηρούνται για να πάψει η διάκριση κατά της Νάση Ντελέη. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ε, ότι ήταν ερευνήτρια πλήρους απασχόλησης και το 2017 το εφετείο ε, ε, απεφάνθη ε, ότι θα πρέπει να τις καταβληθούν οι μισθοί που τις οφείλονται. Αλλά εννιά χρόνια αργότερα το αντίστοιχο τμήμα του ακυρωτικού δικαστηρίου ακύρωσε αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και βεβαίω το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας έδρασε τάχιστα. Το Νοέμβριο του 2017 περίεκοψε το μισθό της να συντελέει κατά θα δείτε στο παράρτημα επίσης ε, ε, τη Γαλλίδα ε, Ισαμπέλ Μορέ που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Το 1993 έπαιρνε 1424 Ιταλικές λιρέτες που ε, και σήμερα παίρνει μισθό λιγότερο, 23 χρόνια αργότερα. Και δεν είναι ε, η μόνη. Προφανώς η διαδικασία της Μπολόνια δεν έχει φτάσει μέχρι το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Θέλω να αποτύσω φόρο τιμής στην κυρία Ντάλιν και τον Σάρτζο Κοφεράτη, ευρωβουλευτές που έκαναν ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Μακρόν, ο κύριος Μακρόν, η κυρία Μέη, ο κύριος Μπαρνιέ και άλλοι ε, δεν μπορούν να επιτρέπουν στην Ιταλία να μην ε, υπακούει στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αν θέλει να επιβιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει κατεπηγόντω να τηρούνται αυτά. Για τι διαπραγματεύσει του Brexit, ο κ. Φερχόφστατ είπε δεν πρόκειται ποτέ να συνενέσουμε εάν δεν έχουν ε, λυθεί με τρόπο ικανοποιητικό τα θέματα των πολιτών. Στι 29 Απριλίου του 2017 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι οι εγγυήσει θα πρέπει να είναι αποτελεσματικέ, εφαρμόσιμε και μη διακριτικέ. Οι πολίτε θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά του με ε, τρόπο απλό χωρίς γραφειοκρατία. Ελπίζω η Επιτροπή σας να πιέσει το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε η Ιταλία ένα κράτος μέλος να πάψει να ε, κάνει διακρίσεις εις βάρος όλων των υπολείπων ε, κρατών μελών και των πολιτών αυτών των κρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ. Η κυρία Ράμου ή ο κύριος Πέρης Φλόρες. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος μου δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ σήμερα. Θα απαντήσω σε, για αυτή την υπόθεση που είναι η παλιότερη υπόθεση που έχουμε όπως υπογραμμίσατε. Ξεκίνησε πριν αρχίσω εγώ να δουλεύω για την Κομισιόν. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Κομισιόν ε, παρακολουθεί πολύ στενά αυτή την υπόθεση. Θα θυμάστε ότι το 2004 η Κομισιόν ε, μείνει την Ιταλία, ε, προσέφηκε κατά της Ιταλίας στο δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε ότι ακόμη και αν η Ιταλία δεν συμμορφωνόταν με παλαιότερη απόφαση, η παραβίαση αυτή έχει σταματήσει. Ε, σημείωσε η Κομισιόν αυτή την απόφαση και έδρασε αναλόγως. Μετά από αυτό, υπενθυμίζω το ιστορικό, διότι καλό είναι να το θυμόμαστε. Μετά από αυτό, είχαμε την νομοθεσία Gemini, που από τη μία πλευρά καθιέρωσε κάποια συγκεκριμένη ερμηνεία της νομοθεσίας ε, για να διθέτει στην κατάσταση και από την άλλη ε, ακύρωσε όλες τις εκκρεμούσεις υποθέσεις στα εθνικά δικαστήρια. Είπε πρέπει να σταματήσουν. Η Κομισιόν εξέθεσε το πρώτο κομμάτι της διακριτικής μεταχείρισης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν αδύνατο να αποδειχθεί διακριτική μεταχείριση, διότι πρέπει να καταλάβετε ότι σε μια διαδικασία παραβάση το βάρος της απόδειξης εναποκτεί στην Κομισιόν. Εμείς λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσαμε ότι δεν υπήρχε παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για αυτό το κομμάτι. Στο άλλο κομμάτι, την πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα, το άρθρο 27, εκεί ξεκίνησε η Κομισιόν ένα διάλογο με τις Ιταλικές Αρχές και όπως ενημερώθηκαμε, όπως ενημερώσαμε αυτή την Επιτροπή τα τελευταία δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κάποιο τρόπο έπεισε τις Ιταλικές Αρχές να υιοθετήσουν ένα, να βρουν μια λύση για αυτό το θέμα. Οι Ιταλικές Αρχές, η Ιταλία υιοθέτησε μια νέα νομοθεσία σας ενημερώσαμε για αυτό το νομοσχέδιο στην τελευταία ανακοίνωση και τώρα που έχει υιοθετηθεί ο νόμος, η Κομισιόν μελετά το νόμο αυτό και θα σας γράψουμε όταν θα έχουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτής της νομοθεσίας. Αυτό είπαμε και την τελευταία φορά. Τη περασμένη φορά ήταν νομοσχέδιο, τώρα έχει ε, περάσει πλέον, έχει εγκριθεί. Ε, αυτά είχα να πω. Θα σας ενημερώσουμε. Άριστα. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν κάποια άλλα μέλη που θα ήθελα να παρέμβουν για το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτό το θέμα σήμερα το πρωί. εσύ βλέπετε καλά θα έχετε καταλάβει ότι δεν είμαι η κυρία Ντάρλεγγ Την αντικαθιστώ γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις στο Λονδίνο σήμερα το πρωί. Κυρία Πρόεδρε, η τελευταία απόφαση του Ιουλίου 2017 του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιταλίας αποτελεί προσβολή μίας από τις ε, τέσσερις ελευθερίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση αυτή και είναι απολύτως απαράδεκτη. Το δικαστήριο έδειξε ότι περιφρονεί τα δικαιώματα των ε, ξένων λεκτορών που πηγαίνουν στην Ιταλία για να συμβαλούν ε, διδάσκοντας ε, στην Ιταλική κοινωνία. Κυρώνοντας αυτή τη διάκριση κατά αυτόν, αυτό δείχνει ότι μετά από 40 χρόνια και 6 υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πραγματικά ε, δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα. Έχω γράψει, έχουν γραφτεί πολλές επιστολές ε, από την ε, Ένωση Ξενών Ελεκτρών της Ιταλίας στον πρόεδρο Γιούνκερ και από τη συναδελφό μου την κυρία Ντάλιν και είναι σαφές ότι δεν υπάρχει βούληση να βρούμε μια λύση για αυτή την κατάφορη παραβίαση του Ευρωπαϊκού Νομοθεσίου αλλά το μόνο που κάνουμε υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα τα συμφέροντα των πανεπιστημίων υποστηρίζοντας αυτή την κατάφορη ε, περιφρόνηση των ε, ξένων λεκτόρων. Ε, σε εποχές όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διασφαλίσει τα δικαιώματα πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν και όταν το Ηνωμένο Βασίλειο φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει ότι είναι αποφασισμένη να προστατεύσει και τα δικαιώματα πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που εργάζονται σε άλλε χώρε. Εύκολα καταλαβαίνει κανεί, γιατί δεν λαμβάνει ισχυρή δράση η Κομισιόν για να ε, διασφαλίσει ε, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Κάτι που θα έπρεπε να κάνει ο σταματοφύλακα των συνθήκων. Και θα ήθελα να προσθέσω και δύο δικά μου λόγια στα όσα μου ζήτησε η κυρία Ντάλεγκ να πω. Ε, όλο αυτό προσβάλλει το τομέα της ακαδημαϊκής ελευθερίας όπου το σύνολο των ακαδημαϊκών ε, συμμετέχουν στη συνολική ακαδημαϊκή γνώση όπως μου είπε ένας πανεπιστημιακός ε, το θέμα δεν είναι ότι εμείς ε, είμαστε στην Ευρώπη για 40 χρόνια είμαστε στην Ευρώπη 900 χρόνια ως πανεπιστήμια και εργαζόμαστε συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε το άθροισμα της ευρωπαϊκής γνώσης το θέμα αυτό θα πρέπει να τεθεί ως επίγον θέμα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Απασχόλησης. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα πρέπει να εξετάσει τα συνταγματικά αποτελέσματα που έχει αυτή η συμπεριφορά των Ιταλικών Δικαστηρίων. Κυρία Πρόεδρε, αυτή η αναφορά που είναι θεμελιώδη σημασία για την Ένωσή μας πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Ε, πολύ επάξια ε, αντικαταστήσατε την κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ και να έρθετε εκπροσωπώντας τον εαυτό σας την άλλη φορά. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Άλλους βουλευτές που θέλουν το λόγο έχουμε. Όχι. Να ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Πέτρη. Θα ήθελα να κάνω μόνο μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτιμώ βέβαια πως το βάρος ευθύνης ε, σε τέτοιες περιπτώσεις το ΔΕΚ ε, βαρύνει την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το καταλαβαίνω και το κατανοώ και νομίζω ότι έχω δείξει πως υπάρχουν πολλές τέτοιε περιπτώσεις. Έχουμε για παράδειγμα αυτή τη συνάδελφο στην Πολόνια που πληρώνεται σήμερα αυτό που πληρωνόταν ε, πριν από 23 χρόνια. Άρα λοιπόν εφόσον υπάρχει αυτό το βουνό αποδεκτικών στοιχείων γιατί πιστεύετε εσείς ότι δεν μπορείτε να τεκμηριώσετε την υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απαντήσει. Δεν μπορώ να προσθέσω πολλά παραπάνω. Ε, σας τα έχουμε στείλει και γραπτός τον Αύγουστο του 2014. Σας στείλαμε στοιχεία για την περίπτωση αυτή διακρίσεων. Το γεγονός πως υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες των δικαστικών αποφάσεων και διαφορετικές ερμηνείες του Ιταλικού δικαίου είναι κάτι το φυσιολογικό. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται στα Ιταλικά δικαστήρια και ο αναφερόμενος το γνωρίζει. Δηλαδή, πολλοί από αυτού τους διδάσκοντες έχουν κερδίσει την υπόθεσή του στο δικαστήριο και κάποιοι άλλοι την έχασαν. Είναι φυσιολογικό. Είναι τα Ιταλικά δικαστήρια που έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν βασιζόμενοι ε, στο Ιταλικό δίκαιο. Fine. That Μάλιστα. Κλείνει η συζήτηση στο σημείο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο θέμα ε, λέγοντας πως η αναφορά αυτή παραμένει ανοιχτή. Διανύουμε την εποχή βέβαια του Brexit και περιμένουμε και μια γραπτή, ενημερωμένη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας την παρουσιάσατε, τη θέλουμε και γραπτά. Και αυτό σε σχέση με το νέο Ιταλικό νόμο. Και προσωπικά θα ήθελα οι συνάδελφοι να στηρίξουν την πρότασή μου που είναι να αναφέρουμε και να παραπέμψουμε, το θέμα αυτό στον Κίφερ Χόσταχτ που είναι ο διαπραγματευτής μας ε, και στην Διευθύνσουσα Επιτροπή για τον Brexit γιατί έχει να κάνει με την κατάσταση και την ελευθερία μετακίνησης και του δικαιώματος των δικαιωμάτων των πολιτών όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Πέτρη. Αν συμφωνείτε μαζί μου μπορούμε να προχωρήσουμε με τον τρόπο αυτό. Πολύ ωραία. Σύμφωνο κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να σας πω πόσο σας εκτιμάμε για, για την αντοχή σας. Έχει πολλά χρόνια αυτή η υπόθεση, αλλά ελπίζω πως κάποια μέρα θα έχουμε θετική κατάληξη και ας κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε για να το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας εύχομαι καλό ταξίδι. Ας πάμε τώρα στην επόμενη ε, αναφορά που είναι η 0906 αφορά την περιβαλλοντική προστασία στην περιοχή του Πιεμόντε στην Ιταλία. Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα γεωργών από την Αυστρία. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ελπίζω να ήρθατε από όλα τα μέρη τη Αυστρία, όχι μόνο από τη Βιέννη. Υπάρχουν λίγοι αγρότε στη Βιέννη, στην πόλη, αλλά να ήρθατε και απ' έξω από τη Βιέννη. Και ελπίζω να δείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα εδώ στις Βρυξέλλες σήμερα. Θα ήθελα μάλιστα να πω ότι τώρα βρίσκεστε στην καρδιά τη Ευρώπη, οπότε προσπαθήστε να αισθανθείτε τον παλμό και ευχαριστείτε τις, ευχαριστηθείτε τις Βρυξέλλες, οι οποίες είναι μια χαρά πόλη και μάλιστα σήμερα δεν βρέχει κιόλας, οπότε ευχαριστηθείτε το γιατί είναι κάτι σπάνιο. Το λόγο έχει ο αναφέρον. Ε, non sta andando avanti il... ξεκινάω τις διαφάνειες. Θα σας δώσουμε κάποια βοήθεια κύριε Κεμέλο. Ah, Thank Καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέα Κεμέλο και είμαι ο Δήμαρχος του Τζομάνο Κεγκαλέζα. Σας ευχαριστώ για το χρόνο. Αφορά ή αναφορά την περιοχή Βαλεντόρα στην Ιταλία, μια περιοχή γεωργική όπου ε, καλλιεργούνται οποροφόρα. Μέσα στις δεκαετίες έχουν αντικαταστήσει ε, τις παραδοσιακές καλλιέργειες διάφορα λατομεία χαλικιού και άμμου. Η Βαλεντόρα θεωρείται από τις σημαντικότερες περιοχές της Ιταλίας για την εξόρυξη ε, τέτοιων υλικών. Ας πάμε θα το διαβάζω κατευθείαν η Βαλεντόρα θεωρείται σημαντική ε, ε, περιοχή για την ανθρώπινη κατανάλωση, για προϊόντα ανθρώπινης κατανάλωσης ε, από, και για τα νερά και εκεί έχουμε πάρα πολλά απόβλητα και βιομηχανικά και ειδικού τύπου και παρότι υπάρχουν υποχρεώσεις να μην υπάρχουν χωματερές εκεί υπάρχουν αυτή τη στιγμή έξι 5 ε, εκατομμύρια κυβικά μέτρα ε, και υπάρχει δίθηση προς τα απόσημα ύδατα. Ωστόσο, προσέξτε, τα υπόγεια ύδατα είναι... θεωρούνται ενιαία. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ε, του, των υπόγειων υδάτων σε μεγάλο βάθος και σε μικρό βάθος. Έτσι λοιπόν σε 100 μέτρα βάθος στα πηγάδια υπάρχουν ε, σήμερα κατάλοιπα παρότι υπάρχουν φίλτρα ενεργού άνθρακα για να διασφαλιστεί ε, ε, το ότι το νερό θα είναι πόσιμο. Από το 2004 συνεχίζεται αυτό και είναι αδύνατον πλέον να εξαλειφθούν οι πηγές ρήπανσης, οι δυνατότητες αποκατάστασης και εξυγένσης θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί. Παρόλα αυτά έχουν δημιουργηθεί και άλλες ε, χωματερές. Ε, ε, Συμπληρώνω αυτές που υπάρχουν. Ο υπουργό Περιβάλλοντος Ιταλίας έχει δηλώσει ότι τα υπόγεια ύδατα κοντά στις χωματερές αυτές θεωρείται μη πόσιμο λόγω των τιμών που έχουν διαπιστωθεί εκεί. Στο Τρατζονα Βερτσελέζε ε, το πηγάδι βρίσκεται μόλις 3 χιλιόμετρα από την χωματερή LC2. Σήμερα λοιπόν παρατηρείτε ότι στο Δήμο αυτό υπάρχει παραβίαση της αρχής της προφύλαξης όπως προβλέπεται από την Ευρώπη και διαπιστώνται πολλές παραβιάσεις της οδηγίας 31 του 99 της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χωματερές βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια ε, βάσει της 3199 ε, ε, αυτή η οδηγία πρέπει να θυμηθούμε ότι επιτρέπει την τεχνητή συμπλήρωση και όχι αντικατάσταση του φυσικού εμποδίου. Σε αυτή την περίπτωση εδώ δεν υπάρχει καθόλου ο κίνδυνος διήθησης των ρήπων λόγω της απουσίας ε, ε, του φυσικού εμποδίου συνεπάγεται και την παραβίαση της οδηγίας 31 Δεύτερον, οι χωματερές βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές, σε ε, ορισμένες περιπτώσεις μερικές δεκάδες μέτρα από γεωργικές περιοχές και από υπογεία ύδατα. Κατάφορη παραβίαση της 31 του 99 η εγκύτητα ε, σε κατοικημένες περιοχές παρεμβαίνει στο άρθρο 8 της 3199. Είναι αδύνατον να, ε, να υπάρχουν χωματέρες κανονικά σε τόσο μικρή απόσταση από κατοικημένε περιοχές. Αυτό που ζητείτε να επελθευτεί η συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Όλες οι χωματέρε που υπάρχουν σήμερα στη Βαλεντόρο ε, παρουσιάζουν τον κίνδυνο διήθηση. Γι' αυτό ζητάμε ε, το μη κλείσιμο της αναφοράς και να αναλυθεί κατά πόσο υπάρχει παραβίαση των ευρωπαϊκών ε, κανόνων. Και δεύτερον, ζητάμε βοήθεια. Ε, ε, ζητήστε εσεί εκ μέρου μα από τι Ιταλικέ Αρχέ να απαγορεύσει την περαιτέρω δημιουργία χωματερών σε αυτέ τι περιοχέ και στα, με, αποτέλεσμα τη ρήπανση των υπογειών Να προσθέσω ότι στις διάφορες εκδρομές που κάνουμε με τα παιδιά των δημοτικών σχολείων, τα παιδιά μας ρωτούν γιατί σε αυτή την περιοχή υπάρχουν τόσες ε, περιοχές υγειονομικής ταφής ε, αφού υπάρχει νερό το οποίο τροφοδοτεί τα πηγάδια, ε, νερό που πίνουμε εμείς και βρίσκεται σε τόσο κοντινή απόσταση από τους χώρους αναπόθεσης απορριμμάτων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thanks to you for your... Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Και προσωπικά Χαίρομαι που έρχεται δήμαρχος της περιοχής. That's, that's very... Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε αυτοπροσώπους. Yes. Uh, and I know that there are some Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την περιοχή του Πεδεμοντίου. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Ε, πραγματικά ε, είμαι βέβαιη ότι είναι καταπληκτική η περιφέρεια αυτή και έχουμε και συναδέλφους εδώ. Ωραία. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρευρίσκεται εκπρόσωπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Thank you, Madam. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ μάλιστα και τους αναφέροντες για την παρουσίασή τους εδώ και για τα έγγραφα που μας παρουσίασαν, τα οποία ήταν πολύ πλήρη για αυτή την αναφορά. Η αναφορά αυτή, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, ε, αφορά την παρουσία πολλών ε, χωρών υγειονομικής ε, απόδοσης απορριμμάτων ε, σε μια περιοχή. Σε μια περιοχή η οποία όπως φαίνεται δεν είναι και ιδανική για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις διότι περιλαμβάνει υπόγεια τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση που δεν διαθέτει φυσικό εμπόδιο όπως είπαμε γεωλογικό και με χωματέρες που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές και γεωργικές περιοχές. Είναι και γεωργική περιοχή αυτή και έχει σημαντικά ε, υπόγεια υδατά. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η διήθηση ε, ρήπων ε, στα υπόγεια υδατά. Και αφού πρόκειται για υδατά τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανθρώπινη κατανάλωση, το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Στην αναφορά αυτή ε, ξαναβλέπουμε κάποιες επικρίσεις που έχουν γίνει κατά της Ιταλίας όσον αφορά τη διαχείριση των χωματερών. Τη διαχείριση και την μετεπιχειρησιακή φάση. Εμείς έχουμε λάβει πολλές ε, ειδοποιήσεις γι' αυτό που αφορούν όλη την Ιταλία από το βορρά μέχρι νότο και η Επιτροπή επ' αυτού πραγματοποιεί μια δράση παρακολούθησης σε πολλά επίπεδα. Έχουμε την εκτέλεση της απόφασης ε, του δικαστηρίου που καταδίκασε την Ιταλία για την παρουσία πολλών εγκαταστάσεων χωματερών παράνομων στην επικρατεία της. Σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν διασφαλίζει την εφαρμογή της απόφασης, δηλαδή επαληθεύει ότι όλες οι χωματερές αυτές ε, μετατρέπονται ώστε να ε, νομοποιηθούν ε, να νομιμοποιηθεί η κατάσταση. Δηλαδή πληρώνει κάποιο πρόστιμο η Ιταλία για αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης έχουμε μια άλλη υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου που αφορούν παραβίαση του άρθρου 14 της οδηγίας για τις χωματερές σε σχέση με χωματερές που ήδη λειτουργούν ή που ήδη έχουν άδεια πριν τεθεί σε ισχύ η οδηγία για τις χωματερές. Εδώ αυτό αφορά περίπου 50 χωματερές που έπρεπε ή να έχουν κλείσει ή να ε, συμμορφωθούν, το οποίο δεν συνέβη και η Ιταλία. Λοιπόν, ε, κλείθηκε να απαντήσει για όλε αυτέ τι στο δικαστήριο. Και επίσης έχουμε διάφορες περιπτώσεις που μας έχουν επισημανθεί λόγω καταγγελιών, αναφορών, γραπτών ερωτημάτων. Ε, αυτή τη στιγμή ελέγχουμε όλε αυτέ τι υποθέσει για να καταλάβουμε αν είναι δομικό το πρόβλημα, αν είναι μεμονωμένε περιπτώσει. Και έτσι θα μπορέσουμε να απολυθεύσουμε κατά πόσο πρόκειται για μια γενική πρακτική συστηματική παραβίαση του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή για μια ε, ε, ε, σποραδική, μια περίπτωση μεμονωμένη. Τώρα για να απαντήσω ε, όσα λέει ο κύριος Δήμαρχος για την κατάσταση στην περιοχή Βαλεντόρα, η Κομισιόν θεωρεί ότι η κατάσταση πράγματι είναι κρίσιμη και χρειάζεται ε, εμβάθυνση. Συμφωνώ λοιπόν, η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και θα πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση, να δούμε τι έχει γίνει, πόσο αποτελεσματικά ήταν τα μέτρα που έχουν εθετηθεί και ενδεχομένως ε, θα πρέπει να δούμε αυτή την κατάσταση στο πλαίσιο των δομικών προβλημάτων ε, που αφορούν τις χωματερές στην Ιταλία, πώς γίνεται η διαχείρισή τους, τόσο κατά τη φάση λειτουργία τους, όσο και στο κλείσιμό τους, γιατί όπως φαίνεται αυτό αποτελεί, δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Ευχαριστώ. Thank you very much and I can assure you that it's not... Ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν συμφωνούν πάντα αναφερόμενος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που συμπίπτουν οι απόψεις Πράγμα που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό. Και θα πρέπει η συγκεκριμένη αναφορά να έχει πάρα πολύ σοβαρή αντιμετώπιση. Οι βουλευτές γιατί δεν ζητούν το λόγο. Α, η κυρία Εύη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Σεσίλια. Ιστορική στιγμή ε, σχεδόν ε, η Κομισιόν ε, ξαφνικά δέχεται όλα αυτά τα οποία επισημαίνει ο αναφέρον, ο Δήμαρχος που βρίσκεται εδώ σήμερα, τον οποίο ευχαριστώ που μας παρουσίασε αυτή την αναφορά. Αναμφίβολα αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και οποίο αφορά την περιοχή αυτή εδώ και πάρα πολύ καιρό και που αφορά και πολιτικές επιλογές ε, εντελώς ε, λανθασμένες και μια επιφανειακή ε, κατανόηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη στιγμή που της επισημάνθηκε αυτό το πρόβλημα. Βλέπω πολύ Βλέπω πολύ θετικά τα όσα είπε η Κομισιόν ε, και θέλω να τονίσω και εγώ κάποια σημεία που υπόθηκαν ήδη αλλά θέλω να τα υπογραμμίσουμε ξανά για περισσότερη σαφήνεια. Έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή που πλήττεται από αυτό το πρόβλημα όχι μόνο το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων αλλά και της ρήπανση του περιβάλλοντος και των υδάτων, ουδάτων που χρησιμοποιούνται ε, για ανθρώπινη κατανάλωση. και διαπιστώθηκε κιόλα ε, από το Κοινοβούλιο πως ε, είναι ανεπαρκής η κατάσταση, ε, ποιότητα των υδάτων ε, λόγω του νικελίου που ε, διαπιστώθηκε εκεί και τι σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων που καταναλώνουν το νερό αυτό. Πέραν της κρίσιμης περιβαλλοντικής κατάστασης, η επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε διαπιστώνει σημαντικά προβλήματα στην περιοχή, διάφορα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να καταλάβουμε ότι το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ιταλία σε περιοχές σαν αυτή πρέπει να αλλάξει. Οι χωματερές δεν αποτελούν λύση για το πρόβλημα των απορριμμάτων. Χαίρομαι φυσικά που υπενθυμίζει η Κομισιόν ότι η Ιταλία δεν ε, πληρεί διάφορους κανόνες και πληρώνει ήδη πρόστιμα για τις ε, χωματερές. Έχουμε ήδη 178 εκατομμύρια ευρώ που έχουν καταβληθεί σε πρόστιμα ε, από τις τσέπες των πολιτών. Ε, δηλαδή οι πολίτες πλέον και χρήματα και με την υγεία τους. Χαίρομαι που αναφέρθηκε επίσης και η νέα έρευνα και η πιθανή προσφυγή στο δικαστήριο και για τις υπάρξεις χωματερές. Αυτό πολύ σωστά επισημαίνει ότι η κατάσταση στην Ιταλία χρήζει περισσότερες προσοχές. Εύχομαι λοιπόν να συνεχίσουμε τις σχετικές αξιολογήσεις της Κομισιόν και φυσικά αυτή η αναφορά θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή ώστε να γίνουν οι έλεγχοι που απαιτούνται στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Κύριο. Τσίριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ έχω εκπλαγεί θετικά. Μετά από τέσσερα χρόνια εδώ στην Επιτροπή Αναφορών είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν δείχνει διαθέσιμη ε, να συμφωνεί, να συνενεί, να συνεχιστεί η έρευνα τέτοιου τύπου με προθυμία και χωρίς την κλασική τους πρόταση που ακούμε σε πολλές αναφορές όπου η Κομισιόν Μα λέει, ναι, έχετε δίκιο επί τη ουσία, αλλά μετά μα λέει, δεν παρατηρούμε καμία παραβίαση ευρωπαϊκή νομοθεσία, οπότε δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αυτή τη φορά, αντιθέτω, η θέση τη είναι διαφορετική. Υπογραμμίζω ότι πραγματικά εκτιμώ το γεγονό ότι η Κομισιόν κατάφερε να υπερβεί την πρώτη τη θέση. Εγώ έχω πάει στο Πιεμόντε, είμαι από εκεί. Ε, έχω συναντηθεί με τον Δήμαρχο και έχω μπορέσει να επιβεβαιώσω και εδώ στην Επιτροπή πόσε χιλιάδε υπογραφέ είχαμε προ υποστήριξη αυτή τη αναφορά. Και εγώ να σα πω ότι η πρώτη φορά που μα έγραψε η Κομισιόν μα είπε μα φαίνεται όλα μια χαρά. Και εκεί είχαμε και μια στιγμή όπου βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση γιατί φάνηκε σαν να επινοούμε εμεί πράγματα ενώ είχαν πιστοποιηθεί επιστημονικά. Και με τα νέα στοιχεία που μας έχουν στείλει τον Αύγουστο, ε, επιτέλους ε, καταφέραμε να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι είναι σημαντικό και ότι η Κομισιόν πρέπει να κάνει κάτι απευθείας από τις Βρυξέλλες. Γιατί αν περιορίζεται η Κομισιόν να λέει ε, στις Ιταλικές αρχές τα πράγματα είναι εντάξει ή όχι, οι ίδιες οι αρχές, ξέρετε, είναι αυτές που έδωσαν την άδεια. Οπότε φυσικά θα σας πούνε ότι τα πράγματα είναι εντάξει. Οπότε πρέπει να πάτε πιο πέρα από αυτό και φυσικά ήμασταν έτοιμοι να μαχηθούμε σήμερα για να ζητήσουμε να παραμένει ανοιχτή η αναφορά αν δεν το είχε πει η Κομισιόν. Αλλά με τη στάση της Κομισιόν τώρα όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Τώρα ζητώ συγγνώμη από τον συναδελφό ε, ε, λυπάμαι που η χώρα μας ε, είναι μάρτυρας τόσων παραβιάσεων αισθάνομαι ντροπή και ενώπιον των άλλων χωρών όπου τα πράγματα αυτά αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Για να κλείσω κυρία Πρόεδρε πρέπει να περάσουμε σε ε, πράξεις. Οι Ιταλικές αρχές πρέπει να λάβουν τη θέση που δεν έχουν λάβει. Και στο τέλος οι πολίτες που δεν φταίνε σε τίποτα πληρώνουν. Διότι όταν η χώρα μας πληρώνει πρόστιμα σημαίνει ότι εγώ ότι πληρώνω το πρόστιμο και οι συγγενείς μου και οι οικογένειες από τη Σικελία ανθρώπων που ζουν χίλια χιλιόμετρα μακριά από εκεί ενώ θα πρέπει να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές της περιοχής. Αντί να επιβάλλουμε κυρώσεις, καλό θα ήταν να παρέμβουμε απευθείας. Ευχαριστώ και πάλι. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αντανόκα, έχετε το λόγο. Thank you. On of the Greens. Θα ήθελα εκ μέρους των Πρασίνων να σας ευχαριστήσω και να εκφράσω και την ικανοποίηση που αισθανόμαστε για μια πολύ επικοδοματική στάση που τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως είναι μια υπόθεση σε εκκρεμότητα, την οποία εμείς προτείνουμε όσον αφορά να διατηρήσουμε ανοιχτή. Εγώ σε προσωπικό επίπεδο θέλω να προσθέσω πως έχω ταξιδέψει πάρα πολύ από το Μιλάνο προς το βορρά κάνοντας σκι. Και έχω περάσει πολύ συχνά από την κοιλάδα αυτή και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα των υδάτων εκεί. Οπότε στηρίζουμε κάθε δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο πάλι στον κύριο Κεμέλο. Εγώ προφανώς είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και εσάς κυρία Πρόεδρε και σας καλώ όπως καλώ και όλους τους ανθρώπους από την ε, Κομισιόν και από τους Ευρωβουλευτές θέλετε να έρθετε να επισκεφτείτε την περιοχή μας ευχαρίστως να σας υποδεχθούμε στην, στο Δήμο του Τρονζάνο γιατί με λίγες εικόνες από ένα βίντεο δεν καταλαβαίνετε την κατάσταση όσο θα την καταλάβετε όπως έχει αντιδείτε πραγματικά. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την επιλογή της. Θα ήθελα εν συντομία να συμφωνήσω με το συμπέρασμα του Αλμπέρτο Τσίριο. Αυτό που ζητάμε εμεί σήμερα από τις Ιταλικές Αρχές και πρώτα απ' όλα από την περιφέρεια του Πιεμόντε, διότι η νομοθεσία για τις κομματερές ε, ε, είναι εξαρτώμενη και από το περιφερειακό επίπεδο, είναι να ε, υλοποιηθούν περιορισμοί όσον αφορά τη δημιουργία περαιτέρω χωματερών και πρέπει να προσέξουμε γιατί τα ύδατα είναι κάτι που, κινείται, που κινούνται. Ε, αυτό το ζητάμε από πολλούς δήμους της περιοχής. Ε, έχουμε συζητήσει με 12 δήμους ε, επί των βασικών αρχών για την ανθρώπινη υγεία όσον αφορά τη χρήση των υδάτων, όσον αφορά τη χρήση των εδαφών και θέλουμε να υλοποιηθούν αυτές οι υποχρεώσεις γιατί Αυτή τη στιγμή πάμε από προσφυγή σε προσφυγή, ε, αλλά με μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με μια επαλήθευση, με κάποια έκκληση, ε, είναι πολύ πιθανό η περιφερεια του Πιεμόντε να μην ε, μας λέει ασάφειε όπως κάνει από τον Αύγουστο και επιτέλους να λάβει μια τελική απόφαση που θα πρέπει να υπάρχει έτοιμη σε κάποιο σιρτάρι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Συνοψίζω. Μην βγάζετε τα ακουστικά σα ακόμα. στην Ευρώπη ξέρουμε ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη για νερό, είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης η διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα πρόβλημα διαρθρωτικό στην Ιταλία και χρειάζεται μεγαλύτερη μελέτη και προσοχή. Βεβαίως, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραμένει ανοιχτή η αναφορά. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα το επόμενο που θα κάνω είναι επίσης ιστορικό και όσοι με γνωρίζετε ε, ξέρετε ότι συνήθως δεν προτείνω διερευνητικές επιτροπές ε, και ε, αντιπροσωπείες γιατί συνήθως δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Εδώ μπορούμε. Λοιπόν, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστούμε και να προετοιμάσουμε μία ε, διερευνητική αποστολή εκεί και βεβαίως ε, θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή και συνεργασία. Θα το προγραμματίσουμε. Βεβαίως. Τι λέτε εσείς κύριε Δήμαρχε, σας αρέσει αυτή η ιδέα. Απολύτως και σας περιμένουμε πολύ γρήγορα και με χαρά ε, να σας υποδεχτούμε γιατί αυτό θα ήταν ένα μήνυμα που θα δείξει ότι η Ευρώπη πέρα από την ομοθεσία και τους κανόνες πραγματικά ε, προσέχει τους πολίτες και τους φροντίζει. Βεβαίως. Συνήθως είναι διήμερες αυτές οι αποστολές που κάνουμε. Αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε και Σαββατοκύριακο εκεί. Ακούω ότι είναι από τις πιο όμορφες γωνιές της Ευρώπης. Μπορούμε να το συνδυάσουμε για να δούμε και την περιοχή σας, ε, Δημαρχέ. Νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παρακαλώ λοιπόν να διαβιβάσετε εκεί στον κόσμο ότι θα το θέσω υπόψη των συντονιστών. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς εδώ και τώρα. Πάντως πολύ στεναρά πιστεύω ότι ενδείκνυται μια τέτοια αποστολή εκεί. Διερευνητική και εξεταστική των πραγμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή. Να προσέχετε την όμορφη περιοχή σας και θα το ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, συνάδελφοι, ελπίζω να είστε ακόμα ε, εδώ μαζί μας. Αγαπητοί συνάδελφοι από τη Μαροκινή Βουλή, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα σας είναι πάρα πολύ σημαντικές από πολλές πλευρές. Ε, το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Κοινοβούλιο είναι από τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και κατοχυρώνεται στις συνθήκες μας. Η Επιτροπή ε, Αναφορών, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, ε, διαδραματίζει ένα πρωταγωνιστικό και όλο ιδιαίτερο ρόλο στην άσκηση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας συνεδριάζουμε μια φορά κάθε μήνα και ε, δίνουμε βήμα στους, βουλευτέ στους ε, πολίτες συγγνώμη, που θεωρούν ότι η νομοθεσία που έχουμε ε, θεσπίσει δεν γίνεται σεβαστή ή εφαρμόζεται με λάθος τρόπο σε κάποιο κράτος μέλος. Και ω μέλη τους Επιτροπή της Επιτροπής έχουμε ως αποστολή να τους ακούμε, να του αφού και να φροντίζουμε στα πλαίσια και εντός των ορίων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων μας τα προβλήματα στα οποία μας εφιστούν την προσοχή να επιλύονται. Γι' αυτό το σκοπό ε, είμαστε σε τακτική και μόνιμη επαφή με τους συναδέλφους που είναι μέλη σε άλλες κοινοβουλευτικέ επιτροπές, καθώς επίσης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι θεματοφύλακα των συνθηκών και δεν διστάζουμε να κάνουμε διαβήματα στις αρχές ε, των κρατών μελών όταν θεωρούμε σκόπιμο και απαραίτητο να τους επιστήσουμε την προσοχή ε, στις καταστάσεις που μας ε, ανησυχούν. Σας ευχόμαστε γόνιμη επίσκεψη και ορισμένοι από εμά θα σας ξαναβρούμε αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας με ιδιαίτερη χαρά. Καλώς ορίσατε. I think, you Νομίζω πως τώρα μπορείτε και εσείς να λάβετε το λόγο και επειδή έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας, εάν ε, θέλετε κάτι να τονίσετε, παρακαλώ είμαστε στη διάθεσή σας. Εάν έχετε κάποια άποψη, κάποια παρατήρηση που θέλετε να κάνετε, μπορούμε να διαθέσουμε κάποιο χρόνο. شكرا السيدة uh, Θέλετε αγγλικά, θέλετε γαλλικά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δέχεστε εδώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι ε, ευρωβουλευτές, είμαστε εδώ για να δούμε πώς ακριβώς γίνεται, πώς παρουσιάζονται οι αναφορές σε εσά, να δούμε πώς θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας γιατί και το δικό μας σύνταγμα προβλέπει τη δυνατότητα κατάθεσης αναφόρων. Και νομίζουμε ότι είναι μια πολύ καλή πρακτική άσκηση για μας, για να μάθουμε από εσάς και να εμπνευστούμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία που μας δείχνετε. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Μπορούμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στην επόμενη αναφορά έτσι ώστε οι μαροκινοί συνάδελφοι να δουν τι κάνουν. Έχουμε τη 1042. Είναι η Friends of the Earth, αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση από την Αυστρία, με 98.500 υπογραφές σχετικά με την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση της ποινιακή ενέργειας που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ και θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπουντίνοβα για να μας πει τα σχετικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να αναφερθεί στην προηγούμενη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Αναφορών το 2014 και να σας παρουσιάσει κάποιες νέες εξελίξεις στο χώρο της πυρηνικής ασφάλειας. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να επαναλάβουμε πως δεν έχουμε την αρμοδιότητα σύμφωνα με το τρέχον νομικό πλαίσιο να λάβουμε δράση να λάβει δράση και να απαιτήσει από τα κράτη-μέλη να καταργήσουν, να κλείσουν τους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί το, ηλεκτρο... το ενεργειακό μείγμα το επιλέγουν ελεύθερα τα κράτη-μέλη. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε πως ε, σύμφωνα με τη νέα οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια, η βασική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια βαρύνει ε, τον κάτοχο της άδειας υπό την εποπτεία του εθνικού ε, ρυθμιστή. Παρ' όλα αυτά, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πυρηνική ασφάλεια παραμένει μια απόλυτη προτεραιότητα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει πως τα κράτη-μέλη που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια να το κάνουν μέσα στο εφαρμοστέο ε, ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας, το οποίο ε, πρόσφατα έχει εμπλουτιστεί και αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε ε, με πολύ προσοχή την μεταφορά του αναθεωρημένου νομοθετικού έργου για την πυρηνική ασφάλεια και θα λάβει δράση για κράτη-μέλη τα οποία δεν συμμορφώνονται στο κομμάτι αυτό. Είναι η πυρηνική ασφάλεια έχει επαναξιολογηθεί και έχουν γίνει μεγάλες αναβαθμίσεις σε επίπεδο ασφάλειας, οι οποίες και συνεχίζονται στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη. Και όλα αυτά απορρέουν από τα stress τεστ, τα τεστ αντοχής που έγιναν μετά τη Φουκουσίμα. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τα υψηλά επίπεδα πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην έκθεση φάνηκε και μια σειρά ε, βελτιώσεων που μπορεί να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και ε, πρέπει να πω πως τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών έχουν αναβυθμιστεί έτσι ώστε να εντάξουν και τις τρέχουσες συστάσεις. Αυτά τα εθνικά σχέδια δράσης πέρασαν δύο αξιολογήσεις από ομολόγους, peer reviews, το 2011 και το 2015, μέσω την ε, ρυθμιστικής ομάδας για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη ε, και παρακολουθήθηκε η εργασία αυτής της Επιτροπής από την, Ευρω... από την Κομισιόν. Στα πλαίσια των Εθνικών Σχεδίων Δράσης τα μέλη αυτής της Επιτροπής ανέλαβαν να παρουσιάζουν μια έκθεση πεπραγμένων ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα και οι πρώτες εκθέσεις, οι περισσότερες, έχουν ε, ληφθεί, ε, ελήφθησαν μέχρι τα τέλη της περασμένης χρονιάς και έχουν αναρτηθεί στο website της Επιτροπής αυτής. Αυτή τη στιγμή οργανώνουμε την πρώτη επίκαιρη αξιολόγηση από ομολόγου στα πλαίσια της αναθεωρημένης οδηγίας για την ασφάλεια με ένα σεμινάριο το οποίο θα οργανωθεί για το μήνα Μάιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει η προσπάθεια αυτή να οδηγήσει σε στοιχεία τα οποία θα πλουτίσουν και θα τροφοδοτήσουν τη συστάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε οι διαχειριστές αυτών των σταθμών να αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια ασφάλεια στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας που διαχειρίζονται. Ευχαριστώ πολύ. Οι συνάδελφοι δεν έχουν λάβει το λόγο. Επιθυμεί κάποιο να σχολιάσει. Όχι. Τότε θα προσπαθήσω να κλείσω το συγκεκριμένο θέμα. Όπως ανέφερε η Κομισιόν, έχουμε και άλλες αναφορές για το ίδιο θέμα. Ωστόσο, αυτή εδώ, όπως είπε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητας, είναι εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών αυτό το θέμα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε αυτή την ε, αναφορά. Βλέπω και κόσμο να γνέφει, ε, συμφωνώντας. Ε, την κλείνουμε λοιπόν και θα στείλουμε μια πλήρη απάντηση στον αναφέροντα για τους σχετικούς λόγους Πάμε στην επόμενη 1403 για την επέκταση του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Τσεχή Δημοκρατία. Δεν ε, παρευρίσκεται ο αναφέρον, αλλά η κυρία Μποχέμοβα βρίσκεται εδώ, οπότε έχετε τον λόγο. Ε, ο συναδελφός σας. Είμαι εδώ για την επόμενη αναφορά αυτή που αφορά το Τεμελίν, ε, το σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, το Τεμελίν της Τσεχική Δημοκρατίας. Δεν έχει εγκριθεί ακόμα, αλλά ο αναφέρον ανησυχεί για το πώς θα, τι θα γίνει με το ε, μελέτη δικτύπου και την σχετική οδηγία. Θέλουμε να δούμε ποιες θα είναι οι πιθανές ε, συνέπειες η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει την πρωτοβουλία το 2014 όπου υπενθύμισε στις τσεχικές αρχές ότι πρέπει να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο της δημιουργίας ένας τέτοιου σταθμού πάνω στο ποτάμι. Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση και η σχετική διαδικασία είναι απαραίτητο να πριν από την τελική έγκριση του έργου να ελεγχθούν οι προηγούμενες ε, ε, μελέτες αντικτύπου. Κάτι που αποτελεί απέτηση και της οδηγίας. Δεν ε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αναμένεται ότι το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το 2025, οπότε είναι αδύνατο σήμερα να προβούμε σε περαιτέρω δράση, αφού δεν υπάρχει κάποια παραβίαση ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι σήμερα. Θα ήθελαν οι συναδέλφοι να παρέμβουν, κύριε Βάιτ. Ε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε. Ε, ε, αξιότιμη εκπρόσωπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευχαριστώ πολύ για την περιγραφή αυτή της αναφοράς. Εκπροσωπώ εδώ τα συμφέροντα των Αυστριακών πολιτών, ανδρών και γυναικών. Όπως γνωρίζετε, η Αυστρία πριν από πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μην έχει πυρηνική ενέργεια και βασικός λόγος ήταν ο ενδεχόμενος κίνδυνος και η απειλή από ατυχήματα για τον ίδιο μας τον πληθυσμό. Αν κοιτάξετε την Αυστρία όμως θα διαπιστώσετε ότι είμαστε περικυκλωμένοι από διάφορα πυρηνικά εργοστάσια πεπαλαιωμένα και σοβιετικού τύπου. Ένα από αυτά είναι το Τέμελιν, το Μπόχουνίτσε και το Πάτς ε, που λέγεται Γκρούσκο σλοβενοκροατικά σύνορα που είναι και σε σεισμογενές ρήγμα επάνω. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να επέμβει άμεσα στο ενεργειακό μείγμα των κρατών μελών. Υπάρχουν όμως διάφορα ζητήματα όπου μπορεί να δώσει την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι γίνεται λοιπόν με την εξασφάλιση, με την προστασία από τα ατυχήματα, τα ενδεχόμενα, τα πυρηνικά. Τι γίνεται με τα ερευνητικά κονδύλια που εξακολουθούν να ρέουν ε, σε αυτό τον κλάδο. Επίσης, τι γίνεται με το εξή ζήτημα πώς ε, προστατεύεται ο πληθυσμός, ε, οι πολίτες σε μια γειτονική χώρα σε περίπτωση ατυχήματος ομιγέννητο. Και ποια είναι το, το ρίσκα. Μπορεί να είναι 1%, μισό της εκατό ή ακόμα και λιγότερο. Να το μειώσουμε τόσο πολύ σε περίπτωση που τελεστεί ένα πυρηνικό ατύχημα. Θα είναι πάντα ολέθριες οι συνέπειες και επιπτώσεις και πέραν των εθνικών συνόρων. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν θα ήθελα να κάνω και μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι η πυρηνική ενέργεια είναι εξοφλημένη. Δηλαδή σιγά σιγά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να φύγουμε από τα πυρηνικά εργοστάσια, να δούμε όσα ακόμα λειτουργούν, πώς θα εγκαταληφθούν. Είμαι υπέρ των ρεαλιστικών λύσεων. Αλλά τώρα να συζητάμε να χτιστούν νέα πυρηνικά εργοστάσια αυτό θα πρέπει να το απαντήσει στεναρά με ένα βροντερό όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί όπως είπαμε οι συνέπειε ενό αντιστοιχήματος είναι τόσο ολέθριε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαπιστώσει ότι σε καμία περίπτωση η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ανανεώσιμη. Για να αποδομηθεί το ουράνιο τραβάμε τα πάνδυνα και από την υγεία και από το περιβάλλον. Και ένα τελευταίο τίθεται και το εξή θέμα. Τι γίνεται με τις επιδοτήσεις που πηγαίνουν εκεί. Πώς μπορεί κάποιος να επιδοτεί ένα τύπο ενέργειας που είναι επικίνδυνο και για τον πληθυσμό αλλά και δεν μπορούμε να αναλάβουμε το κόστος ούτε κατά διάνοια της αποδόμησης των αποβλήτων και την τελική αποθήκευση, τα πυρηνικά απόβλητα αν αυτό το αναλάμβαναν οι εταιρείε, θα ήταν τόσο ακριβή ηλεκτρική ενέργεια από ε, πυρηνικό εργοστάσιο που δεν θα είχε την παραμικρή πιθανότητα και ε, δυνατότητα να ε, ανταγωνιστεί το ρεύμα από άλλε πηγέ και πόσο μάλλον από ανανεώσιμε. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η καρκινοβασία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα έχει φάει τα ψωμιά τη, εν πάση περιπτώσει, η πυρηνική ενέργεια. Είναι πολιτική φύση το ζήτημα, πράγματι. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε να πει κάτι, Όχι. Ωραία. Ας ε, δούμε τι μπορούμε να πούμε ως συμπέρασμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να την θέσουμε σε αναμονή αυτή την αναφορά. Δεν το κάνουμε συνήθως αυτό επίσημα. Απλά δεν θα την ξανανοίξουμε. Εν συντομή θα την διατηρήσουμε ανοιχτή. Θα στείλουμε μια επιστολή στις τσεχικές αρχές για να τους επισημάνουμε το γεγονός ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίε γι' αυτό και θα τους ζητήσουμε κάποια ενημέρωση για το τι σκοπεύουν να κάνουν και για το τι γίνεται με τη σωστή υλοποίηση της ε, οδηγίας περί των υδάτων, ποιες είναι οι προθέσεις τους και όλα αυτά που αναφέρατε εσείς για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Θα τους επισημάνουμε δηλαδή ότι το εξετάζουμε όλο αυτό σε πολύ μεγάλο χρονικό βάθος. Μέχρι το 2025 θα την κρατήσουμε εν αναμονή, δεν θα την ξανανοίξουμε δηλαδή του χρόνου, αλλά θα στείλουμε την επιστολή και θα δούμε τι θα γίνει. Συμφωνείτε? Ωραία. Ευχαριστώ ο κ. Βάιτς την Πρόεδρο. Παρακαλώ, λέει η Πρόεδρο, σα περάσουμε στην επόμενη 956. για τον πυρηνικό σταθμό Τιάνζα 2 ε, που βρίσκεται στο Βέλγιο όπως γνωρίζουμε όλοι. Τρεις χώρες ε, έχουν συνενώσει τις δυνάμεις τους ε, σε μια ομάδα δράσης που ονομάζεται Dryland Region Hange. Ο αναφέρον δεν βρίσκεται εδώ ούτε σε αυτή την περίπτωση αλλά η είναι εδώ, οπότε έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα η Κομισιόν θα ήθελε να τονίσει ότι κατανοεί απόλυτα και παρακολουθεί στενά τις ανησυχίες που εκφράζουν Ευρωπαίοι πολίτες για την ασφάλεια του Τιάνς 2 του πυρηνικού αυτού σταθμού. Ειδικότερα ο Επίτροπος ε, Κλίμα, Κλίματος ε, και Ενέργειας, ο κ. Κανιέτε και οι υπηρεσίες ε, της Κομισιόν Πέρυσης και διάφοροι ενδιαφερόμενοι και εκπρόσωποι των περιφερειακών αρχών και μέλη των κοινοβουλίων των γειτονικών χωρών του Βελγίου καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, οι υπηρεσίες ε, της Κομισιόν παρακολουθούν στενά τα ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας όσον αφορά τα νέα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας ε, συμπεριλαμβανομένου του ΤΙΑΝΣ 2. Ειδικότερα, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή διοργανώνει την πρώτη άσκηση εξέδεση μεταξύ ομοτήμων ε, στο πλαίσιο της σχετικής οδηγίας συμπεριλαμβανομένου του εργαστήριου που θα ε, διοργανωθεί για το Μάιο. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι το Βέλγιο θα συμμετέχει σε αυτή την άσκηση. Το επιλεγμένο θέμα είναι η διαχείριση της γύρανσης των ε, πυρηνικών εργοστασίων. Η Κομισιόν ε, θεωρεί ότι θα βρει σημαντικές πληροφορίες και συστάσεις από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το πυρηνικό σταθμό Τιόνζ και ότι έτσι θα υποστηρίξει τις προσπάθειες των φορέων για περαιτέρω ενίσχυση της πυρηνική ασφαλείας των υπερχόντων εργοστασίων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που, τον οποίο η λειτουργία έχει παραταθεί. Όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια, η Κομισιόν θα ήθελε να τονίσει ότι ενώ η απόφαση για τη μακρόχρονη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, και ενώ η πρωτεύουσα ευθύνη για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών ε, εναπόκειται στους ε, διαχειριστές των πυρηνικών σταθμών, η πυρηνική ασφάλεια και προστασία των πολιτών και φυσικά και του περιβάλλοντος αποτελούν απόλυτες προτεραιότητες για την Κομισιόν. Δεδομένων αυτών, ο ρόλος της Κομισιόν είναι να διασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη που επιλέγουν ε, την πυρηνική ενέργεια θα το πράττουν με πλήρη συμμόρφωση ως προς, το ευρωπαϊκού ως προς το ευρωπαϊκό πλαίσιο πυρηνική ασφάλεια. Έτσι λοιπόν οι υπηρεσίε τη Κομισιόν παρακολουθούν στενά την υλοποίηση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου τη Ευρατόμ συμπεριλαμβανομένη τη τροποποιημένη οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια και θα λάβουν ε, όλε τι απαραίτητε ε, νομικέ δράσει κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τι νέε απαιτήσει. Τέλο, θα ήθελα να πω ότι οι υπηρεσίε της Κομισιόν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι όλες οι σχετικές πληροφορίε και τα σχετικά έγγραφα που ζητούν οι αναφέροντες όσον αφορά το πυρηνικό σταθμό Τιόνς 2 έχουν σταλεί. Το τελευταίο εστάλει τον Νοέμβριο του 2017. Ευχαριστώ. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Η κυρία Σντανόκα. Uh, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι συστάσεις που μόλις προτάθηκαν αξίζει να υποστηριχθούν. Uh, important case. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και παλιά υπόθεση από το 2016 και περιμέναμε πάρα πολύ για να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δράσεις που αναλαμβάνει τώρα. Και ο πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Σούλτς στέλνει διάφορες επιτροπές, επιστολές. Θέλουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση και τις συστάσεις, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να αποσταλεί και στην υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας στην Αυστρία. Okay, so this... Ωραία. Κοιτάξτε, δεν είναι και τόσο παλιά αναφορά αυτή, αλλά είναι τεράστια ε, επί της ουσίας. Και όπως είπαμε, το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η αναθεωρημένη οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια πρόκειται να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Τον Αύγουστο του 2017 έγινε αυτό και η θεωρημένη οδηγία για τις βασικές προδιαγραφές ασφαλείας θα πρέπει να έχει μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο μέχρι το Φλεβάρι του 18. Λοιπόν, θα πρότεινα να κάνουμε το ίδιο με τη συγκεκριμένη αναφορά, να την αφήσουμε ανοιχτή, να στείλουμε επιστολή λέγοντας ότι την παρακολουθούμε και <clears throat> περιμένουμε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιημένη για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Ίσως μετά το εργαστήριο και όταν θα έχετε συνοψίσει και τα αποτελέσματα. Γιατί και αυτό θα ρίξει νέο φως σε όλο αυτό το θέμα. Ωραία. Συμφωνείτε όλοι? Ναι, ναι, θα στείλουμε επιστολή και στους Βέλγους. Στην βελγική κυβέρνηση λέγοντας ότι ενισχύει πάρα πολύ η Επιτροπή μας ε, σύσσωμη και το θέμα της Αυστρίας. ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ε, το έχει υπόψη, το έχει ε, διαβιβαστεί αναφορά, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Το έχουν και το παρακολουθούν, δεν χρειάζεται να το ξαναστείλουμε. Νομίζω αυτό είναι ο καλύτερος ε, δρόμος να ακολουθήσουμε. Ωραία. Πάμε πάλι στην Αυστρία τώρα. Αναφορά 581. Ε, σχετικά με την ενιαία πανευρωπαϊκή ασφάλιση αστικής ευθύνης αποτυχήματα σε πυρηνικούς σταθμούς. Αυτή είναι η 1845, ε, εξ ονόματος της οργάνωσης Atom Stop Oberösterreich, ε, σταματήστε τα πυρηνικά από την Άνω Αυστρία, σχετικά με την αστική ευθύνη από ατυχήματα. Γκαμπριέλ Σβάιγκερ παρευρίσκεται η αναφερόμενη έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Ξανασυζητείτε σήμερα αναφορά μας εδώ στην Επιτροπή και το σημειώνουμε αυτό με χαρά. Είναι πολύ μεγάλη ε, η προσήλωσή σας από το 2013 και το ενδιαφέρον σας, αλλά έχουμε αποκομίσει την εντύπωση ότι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ε, μπορούμε να αναμένουμε περαιτέρω βήματα. Είναι γεγονός όμως ότι την τελευταία τριετία ε, σε θέματα αναλογικής και ενιαίας ανάληψης ειστικής ευθύνης στην Ευρώπη δεν έχει επέλθει καμία σημαντική βελτίωση και κάποιες περιθωριακές βελτιώσεις ακόμα της ασφάλισης ε, δεν είναι σημαντικές ούτε αναλογικές ούτε ενιαίες και δεν θα το φυσβητήσει αυτό κανείς παρόν. Βρισκόμαστε στο 7ο έτος μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα και 32 χρόνια μετά το τεράστιο ατύχημα στο Τσερνομπίλ και ε, στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει το κόστος που μπορεί ε, να μην είναι υπολογίσιμο για ε, πολλά χρόνια. Βεβαίως έχουν χρεοκοπήσει εταιρείε ε, των πυρηνικών ε, σταθμών και ο κρατικός κορβανάς καλείται να καλύψει το κόστος. Και στην περίπτωση του Τσερνομπίλ υπάρχει και η διεθνής κοινότητα δωρητών στην οποία ανήκει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια αυτά τα προηγούμενα θα πρέπει να είναι αυτονόητα και από μόνα τους να συνηγορούν υπέρ μιας υποχρεωτικής δράσης για οποιαδήποτε υπεύθυνη κοινωνία και κοινότητα κρατών για μέτρα ε, προφύλαξης και πρόληψης. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε ε, να είμαστε συνήγοροι των πολιτών μας και να διατηρούμε ανοιχτό σου το θέμα. Ο κόσμος βλέπει ξεκάθαρα με ποιο τρόπο ε, ευνοείται η αμυντική βιομηχανία. Έχουν και οικονομικά πλεονεκτήματα. Για να σας διευκρινίσω, διαβάσω μερικά ε, πόσα λένε οι άνθρωποι υπογράφονται στις αναφορές και τι σκέφτονται για να ε, εγγραφούν και στα πρακτικά σας. Ας πούμε, όταν δεν υπάρχει υποχρεωτική αστική ευθύνη, ε, διαστρεβλώνεται το κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό είναι κρυφές ενισχύσεις κρατικές αν αρχίζαμε να συνυπολογίζουμε το κόστος ε, της ε, ε, αποδόμησης και του καθαρισμού θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και είναι φοβερό που τα ωφέλη τα καρπώνονται ορισμένοι λίγοι ενώ το κόστος το πληρώνουν όλοι. Γιατί το αυτοκίνητό μου πρέπει να το ασφαλίσω εγώ ενώ ε, κάποιο που έχει πυρηνικό εργοστάσιο δεν είναι υποχρεωμένο να ασφαλίζει αυτό το σταθμό για την αστική ευθύνη. Αυτά είναι μόνο σύντομε παραθέσει. Μπορώ να σα αναφέρω ε, ολόκληρα και να σα στείλω μέτρα ολόκληρα ε, γράφων των Ευρωπαίων πολιτών που κατανοούν ότι δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε εμείς ε, ως θέμα η ΜΚΟ και το υπερβάλλουμε και το παρατραβάμε. Ε, Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνουμε στεναρά υπέρ της εφαρμογής αυτής ε, της απέτησης από την πολιτική. Ε, η οργάνωσή μας ε, έχει κάνει και άλλη αναφορά ως ενίσχυση της προηγούμενης που βασίζεται και πάλι σε ε, εκατοντάδες και μάλιστα και σε χιλιάδες ε, υπογραφές. Τα πράγματα είναι σοβαρά κύριε και κύριοι, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Γνωρίζετε ότι το μέλημά μας και το αίτημά μας ε, έχει να κάνει με το ηθικό δίκαιο και παρακαλώ να μας βοηθήσετε να δικαιωθούμε. Ευχαριστώ και πάλι που μου δώσετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο. Thank you very Ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε εδώ, που ταξιδέψατε τόσο μεγάλη απόσταση για να μας διαφωτίσετε περισσότερο για το ζήτημα αυτό. Η Κομισιόν βρίσκεται εδώ, παρακαλώ. Άλλη μια παρέμβαση από εσά ζητώ συγγνώμη που σας εξαντλούμε στην κούραση σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σφάγκερ που είναι αναφερόμενη για την παρουσίαση που μας κάνατε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα θα ήθελε να αναφερθεί στην προηγούμενη συζήτηση που έγινε το 2014 στην Επιτροπή Αναφόρων και να δώσει και κάποιες πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει στην ε, ασφάλιση αστικές ευθύνες για τρίτους ε, και τις ε, σχετικές εξελίξεις. Να σας πω πως για το θέμα της αστικής ευθύνης και την ασφάλιση ε, είχαμε και την πυρηνική ε, ενέργεια το 2014 δεν αναλάβαμε δράση γιατί προκρίναμε μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα το θέμα της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών. Και μας οδήγησε αυτό στην τροπολογία, τη σημαντική τροπολογία της σχετικής οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, την οποία ανέφερα προηγουμένως. Έχουμε επίσης τον κανονισμό του Συμβουλίου που δίνει τα μέγιστα επίπεδα ε, ραδιενέργειας στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές σε περίπτωση ατυχήματος, πυρηνικού ατυχήματος ή εκπομπής πυρηνικής ενέργειας. Όλα αυτά ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες προτεραιότητες Ευρωπαϊκή. Ε, Επιτροπής για ε, την Ενέργεια και στην συνθήκη της Euratom στο άρθρο 98 λέγεται πως τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν να συνάπτονται ασφαλιστήρια συμβόλαια για να καλύπτεται ε, κάθε τύπου κίνδυνος. Όμως τα μέτρα αυτά δεν περιγράφονται με λεπτομέρειες μέχρι σήμερα, μια και προσπάθεια έχει γίνει ε, να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να ε, προς υπογράψουν ε, συμβάσεις που θα επιτρέψουν την ασφάλιση αστική ευθύνη από τρίτα μέρη και σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Στα πλαίσια της Ένωσης Κεφαλαίων, η Ασφαλιστική Ένωση στην Ευρώπη έχει ενισχυθεί μέσω παράγωγου δικαίου που έχει να κάνει με τη συνθήκη και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν στην αρχή της χρονιάς φέτος οι υπηρεσίες κομισιών θα παρουσιάσουν μία νέα μελέτη για το θέμα της ασφάλισης, αστικής ευθύνης από σε πυρηνικούς σταθμούς και θα δώσουμε τη δυνατότητα που έχουν οι ασφαλιστικές αγορές και οι ασφαλιστικές εταιρείες στα κράτη-μέλη της Ευρώπης να ασφαλίζουν τρίτους Πιστεύουμε δε πως η μελέτη αυτή είναι ε, προαπαιτούμενο για να δούμε τι θα πρέπει να γίνεται σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος και πώς μπορούμε να επεκτείνουμε την κάλυψη τρίτων στην περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Και θα δούμε αν υπάρχει και χώρος για να αναλάβουμε προτεραιότητα πιο συγκεκριμένη στο χώρο αυτό. Να δούμε τα ε, ελάχιστα επίπεδα τριτασφάλισης που θα πρέπει να λαμβάνει ένας ε, χειριστή σταθμού πυρηνικής ενέργεια, πυρηνικού σταθμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να θεσπίσουμε ε, τα σωστά ποσοστά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, ο κύριος Μάντελ έχει έρθει, τα μέλη είναι εδώ. Ήθελα να το κάνω σήμερα το απόγευμα, μα μια και είσαστε εδώ και θα έχουμε την παρθενική σας παρουσίαση στην Επιτροπή, μια και έχετε ε, αντικαταστήσει τον κύριο Μπέκερ, με χαρά θα σας ακούσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν συνηθίζεται φαντάζομαι μόλις έρθει κάποιο για πρώτη φορά σε μια κομισιόν να παίρνει το λόγο. Αλλά αφού το ζήτημα φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό για μένα, ήθελα πραγματικά να πάρω το λόγο και να ευχαριστήσω την κυρία Σφάγκερ και όλους τους αναφέροντες που θέτουν αυτό το θέμα και που βρίσκονται μαζί μας στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και η αξία είναι αυτό που λαμβάνεις. Θα το γνωρίζετε φαντάζομαι και έχει νόημα πραγματικά ειδικά όταν αναφερόμαστε στην πυρηνική ενέργεια. Επειδή η ενέργεια ε, που παράγεται με την πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να συγκριθεί με τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή. Οπότε δεν είναι μεγάλη προσδοκία, ούτε υπερβολική προσδοκία το να θέλει κανείς να έχει κάποια σωστή ασφάλιση των πυρηνικών εργοστασίων. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι λυπάμαι πραγματικά που η Βρετανία αναχωρεί από την Ένωσή μας Ε, η παρουσία στιγμή είναι κρίσιμη σημασία, είναι μια ευκαιρία να ε, συντάξουμε από την αρχή όλους τους κινδύνους που υπάρχουν ε, στο πλαίσιο της πυρηνικής ενέργειας επειδή η Βρετανία πάντα υπερασπιζόταν την πυρηνική ενέργεια. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την Επιτροπή να διατηρήσει ανοιχτή αυτή την αναφορά ώστε να έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να παρακολουθούμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστούμε πολύ. Εκτιμάμε ιδιαίτερα που στην πρώτη σας συνεδρία συλλαμβάνετε το λόγο και συμμετέχετε και στη συζήτηση. Πολύ καλά. Άριστα, όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο. Κυρία Βαλίνα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε. Ε, ε, ξέραμε ως νέο μέλος, καλωσόρισες και στην Επιτροπή μας και προσβλέπουμε στη συνεργασία σου που σίγουρα θα είναι σημαντική. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω εγώ του συντάκτη αναφοράς ε, των διαφόρων αναφορών για τη συνεισφορά τους και τις ομιλίες τους. Τι καταλάβαμε και τι είναι ξεκάθαρο ότι πραγματικά ε, υπάρχει μια ευαισθησία και συνειδητοποίηση στους Ευρωπαίους πολίτες για την πυρηνική ενέργεια που δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε εμείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως θα πρέπει να φροντίζει να εφαρμόζονται σωστά οι συνθήκες με μέγιστη διαφάνεια όμως σε όλη την πληροφόρηση και την ενημέρωση που έχει. Αλλά και πέρα από αυτό πέρα από ε, τη σωστή ασφάλιση αστικής ευθύνη, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να ασχολείται με το να πείσει τα κράτη-μέλη να εγκαταλειφθεί η πυρηνική ενέργεια που δεν είναι ούτε ασφαλής ενέργεια ε, ούτε καθαρή γιατί σε αυτές τις μορφές ενέργειας ποντάρει πλέον σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει ε, προς τα εκεί να στραφούμε στις ανανεώσιμες και όχι μόνο το 2030 να φτάσουμε στο 35% ανανεώσιμων και θα ήταν θαυμάσιο να το ξεπεράσουμε και να έχουμε και δεσμευτικούς στόχους κάθε κράτος μέλος ε, ξεχωριστά. Ευχαριστώ πολύ. κύριος Βάιτς. Thank you. I, do not want... Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να επαναλάβω την ομιλία που έκανα προηγουμένως. Επειδή βλέπω ότι έχουμε κοινό συμφέρον, και ε, ενδιαφέρον στην Επιτροπή Αναφορών για αυτά τα θέματα και μάλιστα θα έλεγα και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Θα σας παρακαλούσα και θα σύστηνα να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Και τώρα με χαρά θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Σφάγκερ, ε, τη συντάκτρια της αναφοράς αυτή. Ευχαριστώ πολύ ε, ξανά και για την ε, τοποθέτηση σε εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μόνο που έχω να πω εδώ είναι ότι θα παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά ε, την τάξη μεγέθους, για ποιο ποσό πρόκειται δηλαδή. Και θέλω να σας πω ότι η πρώτη μας αναφορά ζητούσε ασφάλιση της τάξεως των 400 δισεκατομμυρίων. Και αυτό δεν είναι κάτι που κατεβάσαμε από το μυαλό μας, η δική μας ΜΚΟ αλλά η γαλλική ε, υπηρεσία, ο Γαλλικός Οργανισμός Πυρηνικής Ασφάλειας μετά τη Φουκουσίμα έκανε υπολογισμούς για αντίστοιχο ατύχημα στην Ευρώπη και έχει καταλήξει σε ζημίες της τάξεως των 423 δισεκατομμυρίων είναι ρεαλιστικά αυτά και αν θυμηθώ τι έγινε το 2014, ο Επίτροπος Σόιτιγκερ είχε πει ότι αυτά που ζητάνε εδώ πέρα κάποιες ΜΚΟ, τριψήφια νούμερα, είναι πάρα πολύ ανεδαφικά και θεροβάμωνα ε, και θα μπορούσε να είναι πολύ χαμηλότερο το ποσό, διψήφιο δηλαδή, ε, πάντα σε δισεκατομμύρια. Δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση αυτά τα λεφτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ας κάνουμε λοιπόν τα εξής. Ε, θα τη διατηρήσουμε ανοιχτή φυσικά και μετά θα έχουμε και το workshop το Μάιο που ανέφερε και η Κομισιόν όπου θα εξετάσουμε το ίδιο θέμα. Διατηρούμε λοιπόν ανοιχτή την αναφορά αλλά δεν θα πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε δράση για κάποιο καιρό όσον αφορά αυτή την αναφορά. Έχουμε ένα ζήτημα εδώ όπου τόσο η Κομισιόν έχει αναθέσει μελέτη όσο και εμείς έχουμε αναθέσει μελέτη εκ μέρους της Επιτροπής μας μελέτη που θα έχουμε μέχρι τα τέλη του έτους ε, αφορά το θέμα της ευθύνης και των διασυνεριακών επιπτώσεων της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένουμε λοιπόν αυτές τις δύο μελέτες με μεγάλη ανυπομονησία και πριν από αυτές δεν υπάρχει λόγος να αναλαβούμε άλλη δράση πέραν του ότι θα ενημερώσουμε την Επιτροπή Ήτρε για την ύπαρξη αυτής της αναφοράς και για το περιεχόμενό της και ενδεχομένω θα στείλουμε και μια επιστολή για να ευαισθητοποιήσουμε τις αυστριακές αρχές να τους ενημερώσουμε ότι το εξετάζουμε εντάξει θα κάνουμε αυτά ωραία λοιπόν αυτό μας προσφέρει τώρα ένα τεράστιο διάλειμμα για μεσημεριανό πηγαίνετε στους ε, βοηθούς σας και πείτε τους ότι θα έχουν ένα μεγάλο διάλειμμα να χαρούν και εσείς και οι καλεσμένοι σας θα έχετε πάρα πάρα πολύ χρόνο για το μεσημεριανό φαγητό. Θα τα πούμε στις 2.30 το απόγευμα.